Mesdames, Messieurs, bonjour. Allez, on va y aller. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ας ξεκινήσουμε. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης θα θεωρηθεί οθετημένο εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις. Καλημέρα σας. η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 8ης και 9ης Οκτωβρίου και της 5ης Νοεμβρίου επίσης θα θεωρηθούν υιοθετημένα εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν τα λέω. Ε, Βίκτορ, Βίκτορ, ησυχία. Και όλοι οι διάφοροι γραμματείς και σύμβουλοι. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Θα ήθελα να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως το γνωρίζετε, σήμερα είμαστε 3η Δεκεμβρίου 2018 και γιορτάζουμε τη Διεθνή ημέρα των ανθρώπων με αναπηρία. Αυτή η μέρα ορίστηκε ως ε, η μέρα των ανθρώπων με αναπηρία το 1992 από τα Ηνωμένα Έθνη και στόχο έχει να προωθήσει την ευημερία και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Αυτή η μέρα είναι μια ευκαιρία για να συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμαστε ε, όσον αφορά την ιδιαίτερη τους κατάσταση. Το θέμα το φετινό τονίζει την αυτονόμηση των ανθρώπων με αναπηρία για μια ανάπτυξη ισότιμη για όλους, βιώσιμη μέσα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης με τον ορίζοντα του 2030. Το πρόγραμμα αυτό δεσμεύεται να μην αφήσει κανέναν στην άκρη τα άτομα με αναπηρίες ως δικαιούχοι αλλά και ως φορείς αλλαγής μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία προς μια πραγματικά καθολική ανάπτυξη συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου της μείωσης των κινδύνων της αστικής ανάπτυξης. Μετά από αίτημα της δικής μας Επιτροπής, το θεματικό τμήμα προετοίμασε μελέτη που θα βρείτε στην είσοδο της αίθουσας. Αυτή εδώ είναι, σας τη δείχνω. Και Στόχο έχει να εξετάσει εις τα προβλήματα προσβασιμότητας στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επέτρεψε να χαρτογραφήσουμε την προσβασιμότητα στα κράτη-μέλη σε τρεις διαφορετικούς τομείς. Τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, τις τοπικές μεταφορές και τον τουρισμό. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι στο σύνολο η προσβασιμότητα των ε, διαδρομών μακρινών αποστάσεων καλύπτεται αρκετά καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό δείχνει την μεγάλη επιρροή που έχουν ε, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί στην προώθηση της ε, προσβασιμότητας. Αντίθετα, η κατάσταση των τοπικών μεταφορών που ρυθμίζονται διαφορετικά ανάλογα με το κάθε κράτος μέλος ή ακόμα και κάθε πόλη Περιφέρεια είναι ακόμα πολύ ανομοιογενής. Έχουμε μικρά κρατημέλη και μεγάλες πόλεις που γενικά έχουν προχωρήσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο προσβασιμότητας, ενώ κρατημέλη κράτη-μέλη ή περιφέρειες αγροτικές παραμένουν τελείως προσβάσιμες σε θέματα τοπικών μεταφορών. Και αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί με εθνικά μέτρα πολύ πιο συντονισμένα αλλά και σε αυτό το επίπεδο η Ευρώπη οφείλει να δραστηριοποιηθεί και να προωθήσει την αλλαγή. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και της ε, ε, Επιτροπής μας ε, που απέδωσε ένα νέο βραβείο στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Εφιούς Τουρισμού για το οποίο τα κριτήρια προσβασιμότητας μετρούσαν ανάμεσα στα τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης για την ε, επίδοση αυτού του βραβείου. Για θέματα πολιτικής τουρισμού, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζεται στις δράσεις συντονισμού και ενημέρωσης. Οι προσπάθειες ε, που γίνονται για την εναρμόνιση των συστημάτων πληροφορικής για την προσβασιμότητα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατέληξαν σε σπουδαία αποτελέσματα και η οι πηγές ενημέρωσης είναι πολλές και διάφορες. Ωστόσο, είναι σημαντικό για μας να θυμίσουμε ότι στην πλειοψηφία των κρατών και των περιφερειών η προσβασιμότητα των μεταφορών και του τουρισμού έχει σίγουρα βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία 10 με 20 χρόνια αλλά πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται και αυτές οι προσπάθειες δεν είναι ακόμα επαρκείς για παράδειγμα, είναι ακόμα πολύ δύσκολο να εξασφαλίσουμε μια αλυσίδα ταξιδιών χωρίς διακοπή για ένα άνθρωπο ε, με αναπηρία, γιατί όλα αυτά ακόμα δεν είναι επαρκώς εναρμονισμένα. Γι' αυτό το λόγο ε, δε θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που, κατε, που στις 8 ε, Νοεμβρίου ε, συμφώνησαν ε, σε μία πράξη για την εναρμόνιση των νομοθετικών, ρυθμιστικών, διοικητικών μέτρων όσον αφορά τις απαιτήσει για θέματα προσβασιμότητας που θα πρέπει να είναι εφαρμοστέα σε όλες τις υπηρεσίες, όλα τα προϊόντα και η Επιτροπή Μεταφορών συμμετέχει στην νομοθετική διαδικασία και θα δείξει ότι ακριβώς αυτές οι πτυχές δεν θα ξεχαστούν. Δυστυχώς θα πρέπει να ομολογήσω ότι σε θέματα μεταφορών οι τροπολογίες μας υπέρ μιας ε, αυξημένης προσβασιμότητας για τους ανθρώπους ε, με αναπηρία ή τους ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα ε, προσέκρουσαν σε μια σημαντική αντίσταση σε επίπεδο του Συμβουλίου. Και το λέω δυστυχώς αυτό είναι απαράδεκτο, ειδικά όσον αφορά όλες τις ε, πολυτροπικές πλατφόρμες στον τομέα του τουρισμού. Το τελικό κείμενο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Ελπίζω πώς θα διορθώσουν τα πράγματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσωπικά πιστεύω ότι πέρα από την υιοθέτηση αυτής της ε, πράξης, θα πρέπει να αφιερώσουμε πολύ περισσότερα μέσα στην προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να εγγυηθούμε σε κάθε πολίτη μία δίκαιη κινητικότητα, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που ε, έχουν κάποια αναπηρία ή έχουν περιορισμένη δυνατότητα κινητικότητας, όπου και αν βρίσκονται σε ολόκληρη την Ένωση, να έχουν μία πραγματική εύκολη πρόσβαση και αυτόνομη πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταφορών. Ε, ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί ε, αυτό το θέμα εμείς θα το καταστήσουμε προτεραιότητα. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Κύριε Τέιλορ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήμουνα υπεύθυνο για την ε, εισηγητή μάλλον και γνωρίζαμε μεταξύ των σκιώδων εισηγητών ότι οι προτεραιότητε τη Επιτροπής Μεταφορών ήταν να καταστήσουμε υποχρεωτικό και τη διευκόλυνση πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία και με αυτούς που έχουν εγκαιστηριακά θέματα στο χώρο του κτηρίου. Δεν είναι χρήσιμο να έχουμε ένα σύστημα μεταφορά που να μπορεί να το χρησιμοποιεί ο καθένα. Έγινε η πρόταση να συμπεριληφθούν όλα τα είδη τοπι, ε, είδη τοπικής μεταφοράς και δεν μπορούμε επίσης να αγνοήσουμε το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ε, συγκινήθηκε ιδιαίτερα Δεν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό και τελικά έκαναν ένα σχέδιο συμφωνίας Ναι, μπορέσαμε να έχουμε εισιτήρια self-service για κάθε άτομο με αναπηρία. Αλλά αυτό που ήθελε να πετύχει η Επιτροπή μας δεν συμπεριληφθήκε. Και υπάρχουν ομάδες από άτομα με αναπηρία που γράφουν για αυτά τα θέματα και είναι πολύ απογοητευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν που μας δώσετε την ευκαιρία να το θίξουμε το θέμα αυτό. Merci, Monsieur Taylor. Monsieur Wim van de Kamp, vous vouliez rajouter un mot La parole est à vous. Κύριε Βαντεκάμ, θέλετε να προσθέσετε κάτι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την πολιτική συνοχή, όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο θα είναι αυτό για τα, θα είναι αυτό για τα άτομα αναπηρία. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι και επίσης γνωρίζουμε ότι ο αγώνας γίνεται και θα πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Είχαμε ένα παράδειγμα πρόσφατα για τα ε, δικαιώματα των ταξιδιωτών με τρένο. Ε, εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε κάποιες βελτιώσεις. Η ελπίδα μου είναι ότι όλες οι τυπικές αρχές και μη οι κυβερνητικές οργανώσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το κείμενο για περισσότερη χρηματοδότηση και περισσότερη ελευθερία. Θα πρέπει και το Κοινοβούλιο μας να προσέξει να επιλύσουμε το θέμα. Σε κάθε χωριό της Γερμανίας και της Ολλανδίας δεν είναι εύκολο, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουν πρόσβαση στις ε, τοπικές ε, περιφερειακές και κοντινές συγκοινωνίες τα άτομα με αναπηρία. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ χρήσιμη έκθεση. Quel, quel que soit Ευχαριστώ κύριε Βαντερκάμπ. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο οι περιφέρειες, οι πόλεις αλλά και οι υπουργοί μεταφορών οφείλουν να καταστήσουν το θέμα αυτό ε, προτεραιότητα. Θα πρέπει να ξυπνήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε όλο τον κόσμο. Κανένας να μην μείνει στην άκρη, κανένας να μην μένει στο δρόμο. Αυτό θα σταλεί από μένα σε όλους τους υπουργούς μεταφορών από αύριο κιόλας. Συνεχίζουμε. Και περνάμε στην πρόταση κανονισμού. όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Διοντολογίας Περιθεωρήσεων που είναι κομμάτι των ψηφοφοριών. Αλλά για να δούμε εάν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες μας θα δω αν, είμαστε, αν έχουμε απαρτία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ε, τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ για να μετρήσουμε κιόλας πως είστε παρόντες. Πολύ ωραία, είμαστε αρκετοί, έχουμε απαρτία για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε και ξεκινάμε. Τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, αποχές, δεν κατάλαβα, ηλεκτρονικός έλεγχος, ε, ψηφίζουμε παρακαλώ γιατί είναι 47. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, αλλά δεν σηκώσατε τα χέρια σας. Τι είναι, Δευτέρα πρωί? Ε, όχι, και όλες απόγευμα είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 49 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Βλοκ α, υπέρ κατά αποχές δεν κατάλαβα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ηλεκτρονικός έλεγχος τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 5 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 5 μάλιστα άρχεται η ψηφοφορία Ε, εντάξει, άμα δεν με πιστεύετε θα επαληθεύσουμε. Λοιπόν, τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Είχα πει ότι εγκρινόταν. Η 55, τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία Συγγνώμη, μπλοκ Β υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ κατά 74. Τι έγινε, 7 7-4, 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπλοκ σε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 Θέλετε να επαληθεύσουμε. Ωραία λοιπόν, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για τροπολογία 18, άρχεται η ψηφοφορία. Εγώ πιστεύω πως ε, ε, εγκρίθηκε τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές δεν κατάλαβα ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την 26 τέλος ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 29, 27 ε, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου, όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της πληροφορίας. 26 ψήφοι υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνεται η έκθεσή σας. Μπράβο κύριε Ουλή. Περνάμε τώρα Λοιπόν, έχουμε την έκθεση για τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας αεροπλοείας. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Et je ferme le Πέρα της ψηφοφορίας. 30 υπέρ, 0 κατά εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Κιστελόρ για την προστασία των ε, ζώων κατά τη μεταφορά στο, ε, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός και εκτός της Ένωσης. Συμβαστική 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχή, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε ε, παλήθευση για την ε, τροπολογία 5, ψηφίζεται ηλεκτρονικά, της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 2. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στην 19 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στη συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροποποιητική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Τροποποιητική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 6 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο, 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, α, εγκρίνεται. Θα επαληθεύσουμε για την τροπολογία 75, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 19 κατά και απορρίπτεται. Είχατε δίκιο. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στο 78. Υπέρ, κατά, αποχές και εγκρίνεται. Νομίζω θα το επαληθεύσουμε. πέρα τις ψηφοφορίες και νομίζω ότι έχει εγκριθεί. Ναι, εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στην 81 ε, υπέρ, κατά, δεν είναι ξεκάθαρο. Επαληθεύουμε για την τροπολογία 81. Πέρα τις ψηφοφορίες και εγκρίνεται. Τροπολογία, τροπολογία 82. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83. Υπέρ. Μισό λεπτάκι. Για το 83 καταπίπτει. Και άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας 27 υπέρ, κατά 5, μία ψήφος αποχής. Σε εγκρίθηκε η, ε, ε, εγκρίθηκε το, ε, η έκθεσή σας. Συνεχίζουμε με την τελευταία ψηφοφορία για την Ο εισηγητής είναι ο κύριος Σαλίνη αναφορικά με την διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τη μην καταβολή οδικών τελών στην Ένωση. Μόνο ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία άρχεται πέρας ψηφοφορίας Συγχαρητήρια κύριε Σαλίνη. Δεν έχετε ψήφους κατά. Καμία αποχή, καμία ψήφος αποχή. Συγχαρητήρια. Ο κανονισμός εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε με το επόμενο θέμα για την ε, για την έξοδο της, ε, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου από την, την Ένωση. Ο εισηγητής, ε, η εισηγήτρια είμαι εγώ σε αυτή την περίπτωση. Περιμένω θα περιμένω αυτούς που πρέπει να εξέλθουν αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε. Στην έκθεση για την ε, ε, τροποποίηση του κανονισμού η, απο, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεσή μου ε, τροποποιήθηκε. Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής η οποία υιοθέτησε την η οποία υιοθέτησε τα ε, τροποποίηση σε περίπτωση μη συμφωνίας για τον Brexit. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ε, με καλές προθέσεις, ξεκινώντας ε, δηλαδή... Ε, έκανε μία, μία, μία καλή ένα καλό σχόλιο, ο οποίο όμως δεν, δεν, δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προσπάθεια ως προς τον Brexit, έχοντας μια νομοθετική ασπίδα σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία. Με αυτή την ασπίδα θεωρώ, λοιπόν, αυτή την ασπίδα θεωρώ ότι θα είναι μέτρα που θα ε, ε, φυσικά άπτονται του χρηματοδοτικού για να ε, ώστε να διασφαλιστούν τα σύνορα στο κανάλι της Μάχης. Μέτρα τα οποία θα δημιουργήσουν νέες ε, οδούς μεταξύ της Ιρλανδίας και των γειτόνων χωρών και αν αυτό ψηφιστεί θα ήθελα να ε, προταθεί ένα μέτρο δικαιοσύνης μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, εδαφών. Υπήρχαν αρκετές ακροάσεις από την Επιτροπή και αρκετές έρευνες για να δείξουν ότι οι διασυνοριακές ε, οδοί μεταξύ Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας, εφόσον μοιράζονται ένα εξωτερικό, εξωτερικά σύνορα με τη χώρα αυτή, θα υποστούν τις συνέπειες, τις αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση που δεν υπάρξει no deal. Έχουμε ποσοτικοποιήσει αυτή την, ε, αυτό τον αντίκτυπο στην έκθεση No Deal των μεταφορών, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, το μόνο παράδειγμα ε, ότι υπάρχει, θα, αναμένεται άνοδος κατά 5% των εισαγωγών, του, των, του κόστου ε, εισαγωγών και εξαγωγών λόγω της, του νέων συνόρων που μπορούν να δημιουργηθούν ε, στα εμπορεύματα διότι οι θαλάσσιες μεταφορές σήμερα στο 100% Η η διαδρομή καλέ Ντόβερ εκτελείται στο 100% αλλά, δεν, αλλά με καινούργια εξωτερικά σύνορα διακινήθενται σε, σε κίνδυνο πολλές θέσεις εργασίας. Τελευταίο παράδειγμα, ε, γνωρίζουμε ότι θα αυξηθούν οι έλεγχοι στα σύνορα στα 20 χιλιόμετρα στο Καλέ και 20 χιλιόμετρα ουρών στα φορτηγά για δύο λεπτά λοιπόν, αυτό θα επιφέρει δύο λεπτά επιπλέον έλεγχο αναφορτηγό. Και σε αυτή την έκθεση, ε, για να είμαι πιο σαφής, προσπάθ... προσπάθησα να δημιουργήσω νέους οδούς ε, ε, σε μια Ευρώπη των 27, δεδομένων αυτών των αλλαγών, τα γαλλικά ε, λιμάνια θα ε, συμπληρώνουν το, το διάδρομο θα, Βόρειας Θάλασσας και Μεσογείου για να, για να διδρύσουμε τους συνδέσμους με την Ιρλανδία αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα διάθετος διάδρομο από την Ιρλανδία μέσω του Ατλαντικού θα περνάει από τη Βρέστη και ε, θα πρέπει φυσικά να προβλέψουμε νέα χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό των, ε, των λιμανιών αλλά και υποδομές ελέγχου και εισόδου ε, των φορτηγών. Προτείνω λοιπόν ένα τη δημιουργία ενός ταμείου έκτακτου για την προσαρμογή από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ταμείο το οποίο θα μπορέσει ενδεχομένω να αντισταθμίσει τα, τις αρνητικές συνέπειες α, της αποχώρησης, ειδικότερα να προστατεύσει τις πιο ευπαθείς περιοχές. Έχουμε ανάγκη χρόνου και χώρου, αλλά και χρήματα δεν έχουμε πλέον το χρόνο σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία και γι' αυτό το λόγο ε, προσπαθούμε να, ε, να, να εγκριθεί αυτή η έκθεση με, μεγαλύτερη ταχύτητα. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕΠ να, να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ως προς την Όσον αφορά στις ε, υποδομές, ακόμα και αν υπάρχει, ε, ακόμα και αν υπάρχει συμφωνία, θα χρειαστούμε περίπου τρία χρόνια για, την, ε, για τον εξοπλισμό των ε, λιμανιών, αλλά και για την αναβάθμιση προκειμένου να έχουμε νέες σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός είναι ο δικός χάρτης που θα σας παρουσιάσω σήμερα ε, για να ε, δω περίπου ποια είναι η θέση της Επιτροπής, αλλά για να μπορώ να δημιουργήσω έναν οδικό χάρτη που θα ε, είναι ξεκάθαρος και θα μπορέσει να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία. Τώρα, το ρόλο, τον λόγο έχει ο κύριος Μιζογέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ απευθύνομαι στην ε, Πρόεδρο και στην έκθεσή σας. Αυτή η έκθεση που θέλει να τροποποιήσει τον μηχανισμό διασύνδεσης για την Ευρώπη και όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Πώς θα σώσουμε δηλαδή τα λιμάνια από την καταστροφή του Brexit, κυρίως τα βόρεια λιμάνια μας. Παρά την ε, καταπληκτική συμφωνία την οποία κατάφερε ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεών μας, ο κύριος Μπαρνιέ, θα πρέπει να βιαστούμε γιατί μια μια ολόκληρη οικονομία και θέσεις επασχόληση θα υποφέρουν αν δεν επιφέρουμε γρήγορα αλλαγέ μέχρι το Μάρτιο δηλαδή του 19 στα, ε, στους θαλάσσιους ε, δρόμους ε, και διαδρόμους η περίοδος μέχρι το 2020 θα χαθεί για τους ναυτικούς μας, τα λιμάνια μας, τους εργαζόμενους τα ντόξ και αν δεν μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τη σύνδεση της Ένωσης με την Ιρλανδία. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδείξει ότι η Ευρώπη χρησιμεύει, ότι ξέρει να εξυπηρετεί και ότι το Brexit είναι μια ευκαιρία να συσφίξουμε δεσμούς και όχι να απομονωθούμε. αντί να αναθέσουμε στους, ε, ε, στο Συμβούλιο μόνο του να αντιμετωπίσει την, την κατάσταση αυτή. Όμως ε, η πρόταση της Κομισιόν δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις που έχουν γίνει από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα λιμάνια, τις ενώσεις, τους προέδρους, των, τους περιφερειάρχες. Η Κομισιόν δεν έχει κάνει μελέτη αντικτύπου και δεν έχει λάβει υπόψη τις διάφορες απόψεις που διατυπώθηκαν στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Επειδή θέλησε λοιπόν να κάνει τα πράγματα βιαστικά και όχι αποτελεσματικά, η Κομισιόν ε, έδωσε ένα ε, μια ημιτελή πρόταση που θα είναι καταστροφική για το σύνολο των γαλλικών ε, λιμανιών και για την οικονομία του, των περιοχών αυτών. Είναι τρελό να αποκλειστούν, αποκλειστούν όλα αυτά τα λιμάνια από τις νέες ρότες, ενώ η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Γαλλία δείχνει μια προφανή σύνδεση ε, ένα πρώτο παράδειγμα που θα αρκέσει νομίζω τα τονάζ ε, οδικών μεταφορών ανάμεσα στην Ελλανδία και τη Γαλλία ήταν ήδη ανώτερα από την, τα οδικά τονάζ ανάμεσα στη, στο Βέλγιο και τις κάτω χώρες το 2017. Γιατί λοιπόν να συμπεριληφθούν μόνο οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί ε, στις νέες διαδρομές αποκλείοντας τα γαλλικά ε, λιμάνια. Θα είναι καταστροφική αυτή η κατάσταση. Συγχαίρω λοιπόν ε, την εισηγήτρια για τις προτάσεις τροπολογιών της και τη στηρίζω στην αποφασιστικότητά της. Η πρόταση τροπολογιών του ΕΛΚΑ θα ε, ε, υποβάλουμε και εμείς για να ξαναμπούν στους, στους διαδρόμους ε, Βόρειας Θάλασσας και Μεσογείου και τα μεγάλα γαλλικά λιμάνια της Βόρειας Θάλασσας και τροποποίηση δεν θέλουμε του, διαδρόμου, του Ατλαντικού διαδρόμου για να ενταχθεί εκεί η Ιρλανδία. Αυτά στηρίζονται πλήρως από την Επιτροπή μας, την Κοινοβουλευτική ε, και ε, βασίζομαι στη δική σας συνεργασία ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα λιμάνια για την ανταγωνιστικότητά τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιζελιέ. Η κυρία... Η κυρία Κριστίνη Ριβονταλόν, μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπω ε, και εγώ έχω σκέψεις που συμφωνούν μαζί σας και μαζί και με τον κύριο Μουζελιέ. Παρότι υπήρξαν ε, ε, διάφορες αντιρρήσεις όταν προτάθηκε αυτό το σχέδιο τον περασμένο Αύγουστο. Το θέμα της προετοιμασίας των λιμονιών σε περίπτωση μη ε, συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια τεράστια πρόκληση που δεν μπορεί να γίνει και να αντιμετωπιστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις. Η, η Κομισιόν έκανε ένα πολιτικής σε σφάλμα επειδή ακολούθησε μόνο μια τεχνική προσέγγιση και σωμάτωσε τα και τα λιμάνια του κεντρικού δικτύου που ήταν ήδη στους διαδρόμους Μεσογείου και βόρεια Θάλασσας, ε, αφήνοντας απ' έξω τη σύνδεση μεταξύ ε, Γαλλίας και Ιρλανδίας και κυρίως της Βρετάνης. Η Κομισιόν μιλά για λιμάνια του γενικού ε, δικτύου όπως η Βρέστη, όμως θεωρώ ότι λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που θα αποτελούσε μία έξοδος άνευ συμφωνίας του της Βρετανίας. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν μια νομική διατύπωση ώστε να υπάρξουν, να υπάρξουν εξαιρέξεις. Θα ήταν δυνατόν δηλαδή να σωματωθεί ένα δίκτυο του γενικού, ένα λιμάνι συγγνώμη, του γενικού δικτύου στο κεντρικό δίκτυο. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν θα ε, επιδείξει νομική εφευρετικότητα προκειμένου να ε, καλυφθούν και αυτά τα λιμάνια. Ε, ο στόχος είναι λοιπόν πολιτικό και εντάσσεται σε μια γεωγραφική διάσταση που καθιστά τις περιοχές της Βόρειας Γαλλίας σημεία εισόδου τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν όσον αφορά τη σύνδεση με, της Ιρλανδίας με την υπηρετική Ευρώπη. Ε, μπορεί να φαίνεται ότι προχωρούμε προς συμφωνία, όμως για την ώρα τίποτα δεν είναι εγγυημένο και θυμίζω πως και όλα τα κοινοβούλια θα χρειαστεί να επικυρώσουν τη συμφωνία αποχώρησης. Γι' αυτό και θα πρέπει να προβλέψουμε, να προετοιμαστούμε για κάθε ενδεχόμενο και ε, δηλαδή για μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία και ε, μπορείτε να βασιστείτε στην ομάδα των σοσιαλιστών για να δουλέψουμε γρήγορα και σας ευχαριστώ για την αρχική σας εισήγηση. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ρεβό Νταλόν. Κύριε Λούντγκρεν, δεν θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι. Ο κύριος Δομινίκ Ρικέ. Ο... Χοροδία γαλλογαλλική. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί βέβαια, αλλά δεν θα επαναλάβω όλα αυτά που υπόθηκαν. Ε, Σημερίζομαι τα όσα είπε η συγγήτρια και οι συνάδελφοι σχεδόν κατά λέξη. Θα κάνω κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι εδώ Αντίθετα με το ότι συμβαίνει εν γέννη, δεν θέλουμε να στηρίξουμε μόνο κάποιες υποδομές μεταφορών και να θυμίσω ότι οι θαλάσσιοι διάδρομοι δεν αποφασίζονται από τον δημόσιο τομέα, αλλά από τους ιδιώτες φορείς και το σφάλμα της Κομισιόν, γιατί είναι λάθος αυτό, θα πρέπει να το κατανοήσουμε, στην ουσία στηρίζει τις υπάρχουσες ε, ε, ε, ρότες και συνδέσεις. Για την ώρα δεν υπήρχαν ε, τέτοιου είδους συνδέσεις για τα γαλλικά ε, λιμάνια γιατί απλούστατα περούσαν, περνούσαν τα πάντα με ρορό από το ε, καλέ. Η στήριξη που μπορούμε να κάνουμε θα είναι η στήριξη στις ε, λιμενικές υποδομές από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν συνδέσεις που δεν υπήρχαν πριν εκτός από τον Ατλαντικό διάδρομο που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν για το Καλέ, ούτε για το Αύγα όμως. Θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν και κατανοούμε γιατί ε, διέπραξε αυτό το πολιτικό σφάλμα η Κομισιόν, το είπε κάποιος ήδη, ίσως αυτό το έκανε για να ξυπνήσει τους Γάλλους, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να γνωρίζουμε και τη φύση της εν λόγω παρέμβασης. Αυτό που επίσης είναι μάλλον σημαντικό εδώ είναι ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα ε, για να λειτουργήσουν ε, οι ε, φορείς διαχείρισης των λιμανιών και οι φορείς διαχείρισης των εμπορευμάτων στα λιμάνια. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω πως είχατε μια πολύ πλήρη έκθεση, όμως αυτό που με εντυπωσίασε ήταν κάτι αυτή η ειδική προσπάθεια. Δεν είναι κακή ιδέα σας, αλλά Πρόκειται για ένα ειδικό ταμείο, το οποίο ξέρουμε τι σημαίνει σε δημοσιονομικό επίπεδο. Εάν πρέπει να προβλεφθεί ένα ειδικό ταμείο και ειδικά ταμεία προσαρμογή στο Brexit ακολουθούμε μια δημοσιονομική προσέγγιση που θα είναι πολύ πιο περίπλοκη από την πρόταση αυτή της αρχικής έκθεσης. Για μένα ήταν αρκετά συναρπαστικό, αλλά πιστεύω πως αυτό θα θέσει διάφορες δυσκολίες. Ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε, να διαβουλευτούμε για να δούμε αν όντως θα πρέπει να ε, κάνουμε αυτή την πρόταση αν θα αντιμετωπίσουμε πραγματικές, ε, ε, πρακτικές δυσκολίες. Έπειτα υπόθηκε ήδη πως η Κομισιόν μας έχει υποβάλει και έχει ψηφίσει και εγώ ο ίδιος υπέβαλα προτάσεις τέτοιες για να μπει το σύνολο των διαδρόμων της Μεσογείου και του Ατλαντικού στον προϋπολογισμό, αλλά ήταν πολύ σημαντικό να ενσωματωθούν σε αυτό το διορθωτικό για το πρώτο τον πρώτο διευθυντικό προϋπολογισμό. Εμείς θα ψηφίσουμε μαζί σας για το θέμα λοιπόν. Είναι αλήθεια πως η Κομισιόν ήταν κάπως αφηρημένη Ε, θα έπρεπε λοιπόν εδώ να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα. Είμαστε σχετικά ομόφωνοι. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Κυρία Κούν. Α, συγγνώμη, όχι, όχι. Διορθώνει η πρόεδρος. Πρώτα ο κύριος Κράμερ. Α, ναι. Επειδή είμαστε ε, από, την ίδια ομάδα, πρέπει πρώτα να μιλήσει η, η κυρία Κούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την έκθεση. Αναφερθήκατε στην Ιρλανδία και βρισκόμαστε στον διάδρομο Βόρειας Θάλασσας Μεσογείου. Το 95% των εμπορευμάτων περνάνε από το Ηνωμένο Βασίλειο και από το Καλέ που είναι το πιο σύντομο πέρασμα 17 ώρες χρειάζεται από την ε, ακτή της Ιρλανδίας μέχρι την υπηρετική Ευρώπη. Είναι πολύ αποδοτική λοιπόν αυτή η οδός και δεν υπάρχει ευβολή ότι ανησυχούμε για το τι θα συμβεί σε περίπτωση ε, εξόδου Brexit χωρίς συμφωνία. Φυσικά και στους λιμένες ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δεσμούς με άλλους ε, λιμένες, να βρούμε εναλλακτικέ ε, οδούς. Μία περίπτωση είναι ο διάδρομος του Ατλαντικού, μία εναλλακτική για την πρόσβαση στον Νότο και στην Ισπανία. Θεωρώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την έκθεση της του Αυγούστου για το πώς μπορούμε να συνδέσουμε τους λιμένες. Όμως τι θα γίνει και με τα λιμάνια στην Γαλλία. Υπάρχει μεγάλη ροή εμπορευμάτων και προ τα εκεί. Όπως και να έχει, Χαιρετίζω την πρότασή σας. Συνεργαζόμαστε στενά με τους σκιώδες συγητές. και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια, δεν πρέπει να περιοριστούμε σε μία πρόταση, μία λύση, γιατί όπως ήδη υπόθηκε υπάρχουν πολλές εναλλακτικές θα αποφασιστούν από τον διεκτικό τομέα εφόσον πρόκειται για εμπορευματικέ ε, μεταφορέ. Όμω υπάρχουν δυνατέ ε, συνδέσει και με την ε, Βορειοδυτική Γαλλία. Ευχαριστώ για την πρότασή σα. Merci beaucoup, Madame Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κλούν. Και τώρα ο κύριο Κράμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω την εκθέση σας, όμως όλα αυτά είναι υποθέσεις. Τι δεν ξέρουμε αν στις 11 Δεκεμβρίου θα, πω, τι θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο μάλλον στο Λονδίνο. Άρα όλα αυτά είναι εικασίες. Ανεξάρτητα κάνουμε λόγους, λόγο για όλα αυτά τα θέματα και διάβασα πρόσφατα ότι ε, θα εγκαταλείψει τους ε, αρμόδιους οργανισμούς του Ενωμένου Βασίλειο και την ΕΑΖΑ. Ισχύει αυτό. Ε, πράγματι υπάρχει αυτή η περίπτωση. Γιατί οι επιπτώσεις ήταν τεράστιες αν δεν θα ανήκει πλέον το Ηνωμένο Βασιλείο στους οργανισμούς αυτούς τους ευρωπαϊκούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για, για το σχόλιο σας. Τώρα θα επιστρέψω στην Επιτροπή και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κόλσον από την DG Move. Ο λόγος ε, είναι δικό σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι η έκθεσή σας ε, τονίζει αρκετά μέτρα που πρέπει να ληφθούν ε, μέσω της νομικής οδού αναφορικά με το θέμα του Brexit και πρέπει να πω ότι εν γέννη συμφωνούμε με τα περισσότερα από τα μέτρα που εσείς θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα. Ωστόσο, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο που προτείνετε εσείς. Η πρόταση που υποβλήθηκε ε, στόχευε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, κάποια μέτρα έκτακτης ανάγκη. Ποια μέτρα έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ε, ε, ληφθούν σε περίπτωση που ε, δεν υπάρχει... δεν υπάρχει συμφωνία με το, με, με το, για το Brexit και σχετικότερα με την, με, με την προστασία της Ιρλανδίας. Προτείνεται λοιπόν ένα πολύ στενό χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2020. Τα μέτρα σας λοιπόν στοχεύουν μόνο στο διάδρομο Ιρλανδίας και Μεσογείου, ο οποίο ο διάδρομος σε περίπτωση Brexit θα κοβόταν στα δύο χωρίς να υπάρχει σύνδεσμο μεταξύ Ιρλανδίας και της υπηρετικής Ευρώπης, όπως συμβαίνει δηλαδή με την Μάλτα ή με την Κύπρο. Και γι' αυτό το λόγο εμείς προβλέψαμε σε αυτή την υπόθεση και μόνο σε αυτή την υπόθεση να επαναδημιουργήσουμε αυτό τον δεσμό με τα τρία λιμάνια που, έχουν το σημαντικότερο βάρος ε, μεταφορών αυτή τη στιγμή και την Ιρλανδία. Και ε, έρχομαι τώρα στις τροποποιήσεις σας. Ε, όσον αφορά στις, στην τροπολογία 10 και 11, η Επιτροπή δεν έχει καμία αντίρρηση να, να προσθεθεί το Καλέ και η Δουνκέρκη στον κατάλογο των τριών ε, λιμανιών ε, του διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας Μεσογείου που θα έχουν και άμεση, άμεση, σύνδεση, με την Ιρλανδία. Ωστόσο, η τροποποίηση των υπαρχουσών διαδρομών με την προσθήκη του Παρισιού ή της Χαύρης ή την προσθήκη της Ιρλανδίας στον Ατλαντικό διάδρομο επιφέρουν επιπλέον μέτρα τα οποία όμως θα πρέπει να είναι μόνιμα και δεν θα σταματάνε 31 Δεκεμβρίου 2020 και θα πρέπει να έχουν σαφή θέση στο, στην αναθεώρηση του ήδη υπάρχοντος πλαισίου. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν καταθέσει προτάσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση ε, που ασχολούνται με την ουσία των, ε, των, ε, των τροπολογιών και τις υποστηρίζουν πλήρως. Όσον αφορά ε, το, το να τεθούν τα λιμάνια στο γενικό ε, δίκτυο, αυτό δεν είναι εφικτό, διότι μόνο τα λιμάνια του κεντρικού ε, δικτύου μπορούν να, να, να, να βρίσκονται και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει και ένας άλλος κανονισμός, ε, ο οποίος θα πρέπει μέσω τροπολογίας να ε, αλλάξει. Επομένως, στο πλαίσιο της ε, αναθεώρησης ΑΧΤΕΟΤΕ θα μπορούσε να ξεκινήσει αυτή η ερώτηση και η Επιτροπή ρωτά τι σκοπεύει, σε τι σκοπεύει αυτή η τροπολογία. Υπάρχουν ωστόσο και ανησυχίες ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί μακροπρόθεσμο και αυτή τη στιγμή ίσως θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τα, για τα πλοία, για, συγγνώμη, για τα λιμάνια του γενικού δικτύου όπως η η το Ροσκόφ. η Κομισιόν συμφωνεί με την πρωτοβουλία του, με του Προεδρείου του Συμβουλίου για τα, ε, για τα λιμάνια και τη χρηματοδότηση του 30%. Κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι στιγμής. Είναι ένα στοιχείο, σημαντικό στοιχείο μέχρι την αναθεώρηση του ΕΧΤΕΟΤΕ, κάτι, ε, κάτι το νέο και νομίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, κάποια, δηλαδή πρωτοβουλία που ήδη έχει υποστηρίξει η, η Επιτροπή μέχρι στιγμής. Όσον αφορά την τροπολογία 6 και 8 για, την, ε, για, τις, για τους ελέγχους στα σύνορα που θα είναι ε, απαραίτητα στον τομέα των τελωνίων, στον τομέα της αστυνομίας, η Επιτροπή από μεθαύριο, σε 6 Δεκεμβρίου, θα δημοσιεύσει στο πλαίσιο του ΕΜΙΟ μία επίκληση προτάσεων για τη χρηματοδότηση των λιμανιών του Γενικού Δικτύου. Επομένω, από την Τετάρτη θα υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθούν ε, με πολύ συγκεκριμένο σκοπό 65 εκατομμύρια, να διατεθούν δηλαδή 65 εκατομμύρια ευρώ για αυτούς τους σκοπούς. Και μέσω από αυτή την, την υποβολή μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα που θα επιτρέψουν στα λιμάνια, όπως για παράδειγμα το, στα λιμάνια της Βρέστης και του Ροσκόφ, να, να προτείνουν ορισμένα μέτρα για την προετοιμασία τους σε περίπτωση ε, μετά το Brexit. Θα υπάρχει λοιπόν ε, μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 6 Δεκεμβρίου και έπειτα. Όσον αφορά στην ε, νέα αναθεώρηση του ΕΜΙΟ, η Προεδρία του Συμβουλίου προτείνει ε, να γίνουν οι χρηματοδοτήσει για τα τελωνία και την αστυνομία αλλά και το τομέα των ε, φυτοϊγειονομικών προϊόντων στο 50%. Η Επιτροπή είναι υπέρ και νομίζουμε ότι ε, θα υπάρξει μια ε, ε, συμφωνία επίσης από το Κοινοβούλιο. Αντιθέτως, αυτή η χρηματοδότηση, εάν τοποθετηθεί σε πολιετές πλαίσιο, δεν, δεν είναι εφικτή λοιπόν κάποια τέτοια, γιατί δεν υπάρχει πολιετές πλαίσιο, ακριβώς γιατί δεν, θα, δεν, θα, δεν υπάρχει προπολογισμό μέχρι αυτή τη στιγμή. Ε, δεν είμαστε απόλυτα υπέρ ε, για ένα επιπρόσθετο έκτακτο ταμείο, ε, διότι αυτό νομίζουμε ότι θα φέρει αρκετά προβλήματα στην πολιτική ανταγωνισμού. Εν κατακλείδη, κυρία Πρόεδρε, είμαστε σύμφωνοι όσον αφορά ε, στην πρόταση της, ε, ε, της προσθήκης της Δουνκέρκης και του Καλέ. Λέμε ναι στην επέκταση των διαδρόμων με μόνιμο τρόπο του μελλοντικού ημιού. Λέμε ναι στην ανάγνωση, στη συγκεκριμένη ανάγνωση των λιμανιών, περιμένοντας εν αναμονή δηλαδή την μεταρρύθμιση ΑΧΤΕΟΤΕ και λέμε ναι στην εκδήλωση ενδιαφέροντος των χρηματοδοτήσεων για τα λιμάνια γενικού ενδιαφέροντος, κάτι που θα επιτρέψει τα λιμάνια να προετοιμαστούν επαρκώς για τον Brexit και λέμε ναι σε, μια, σε τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις στο μελλοντικό εμειό το το μόνο πρόβλημα στο οποίο έχουμε ένα μικρό πρόβλημα είναι στο έκτακτο ταμείο. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που με ακρηγόρησα, αλλά ήταν ένα σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε για την ενθάρρυνσή σας ε, όσον αφορά σε αυτή την εισήγηση. Εάν αυτή η έκθεση τροποποιηθεί, ε, τότε μιλάμε για μια μεγάλη πρόοδο, ε, την προσθήκη δηλαδή των διασυνοριακών λιμανιών στο γενικό δίκτυο. Ε, το κάτι που δεν είχε προβλεφθεί από την Επιτροπή, ωστόσο το Κοινοβούλιο βρίσκεται εδώ. Το δεύτερο πράγμα πρέπει να δείξουμε σε... Ε, είναι ότι θα πρέπει να πω ότι αναφορικά με το ζήτημα του Brexit, οι διατάξεις που σχετίζονται με το Brexit δεν είναι μόνο τεχνικές. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Είναι εξίσου πολιτικές όσο και τεχνικές. Και όταν ζούμε σε μια ατελή κατάσταση που όλα εφευρίσκονται για την προστασία των ε, των, ε, των Ευρωπαίων πολιτών και αυτό είναι μια πολιτική διάταξη, δεν είναι τεχνική η πτυχία αυτή του προβλήματος, είναι πολιτική. Το δεύτερο σημείο κατά είναι πως έχετε μια ε, αρκετά αρκετά τεχνική και αρκετά περιοριστική όψη για τα πράγματα, άποψη για τα πράγματα, που έρχεται σε αντίθεση με το ρόλο μας ως ε, κοινοβούλιο και ως πολιτικούς εκπροσώπους. Και για μένα είναι απόλυτα θεμητό στο, να υπάρξουν ε, τροποποίησεις που ανοίγουν μια πολιτική συζήτηση ε, όσον αφορά ε, την ε, διασύνδεση και ότι αυτά θα είναι και ισχυρά εργαλεία για την προετοιμασία των μεταφορών σε μια μετά Brexit εποχή. Αλλά όχι μόνο στον τομέα των μεταφορών. Ε, στα λιμάνια υπάρχουν και θέσει εργασίας και οι, οι συνέπειες θα είναι μεγάλες αν, ε, αν υπάρξει μια νέα ρότα, ένα νέο διάδρομο. διάδρομος. είναι σκοπός της δικής μας δουλειάς ως Κοινοβούλιο και οι πολιτικές αλλά και ε, νομικές διατάξεις θα αποτελέσουν ε, αντικείμενο συζήτησης ε, μεταξύ των ε, θεσμών. Αλλά χαίρομαι που η Επιτροπή τίνει το χέρι προς τα εμάς. Θα ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε από κοινού. Εμείς είμαστε εδώ για να προβλέψουμε τις συνέπειες. Μου είπατε μου αναφέρατε μια ημερομηνία πριν το Δεκέμβριο του 2020. Πρέπει να προσέξετε, διότι ε, όταν μιλάμε για τους διαδρόμους, ε, αυτό δεν σταματά το 2020. Ξέρετε γιατί. Διότι απλά έχουμε υιοθετήσει τον, ε, το μηχανισμό διασύνδεσης 2 και αυτό εντάσσεται στη νέα πρόταση. Και το Κοινοβούλιο, όπως και η Επιτροπή Μεταφορών, γνωρίζει ε, να γνωρίζει και δεν, το έχει, δεν έχει θέσει ε, το, τη, τη λήξη του στο 2020. Ε, εμείς πρέπει να δούμε τι γίνεται μετά το 2020. Καθώς λοιπόν εντάσσονται στο πλαίσιο της διασύνδεσης, ένα άλλο ζήτημα στο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω, υπάρχουν κάποιοι μοχλοί στους οποίους η Επιτροπή δεν έχει αναφερθεί, που Δηλαδή μιλάμε για, τις, ε, ε, για, την, προ, για την προστίκη, για τη συγγνώμη τροποποίηση ενός έκτακτου ταμείου, γιατί αύριο οι συνέπειες του Brexit ε, για τις περιοχές, για τις, για τις περιφέρειες μπορεί να είναι, μπορεί να είναι δραματικές. Για την Ορμανδία, για παράδειγμα, τότε ποιος θα χρηματοδοτήσει. Αυτό το ταμείο θα πρέπει να μπορεί να, μπορεί να σταθεί αρρωγός. Οι περιφέρειες δεν ζήτησαν τον Brexit, όμως αυτές θα το πληρώσουν το λογαριασμό. Και εμείς πρέπει να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων, ε, ακριβώς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις, περιφέ... περιφέρειες. Και επανέρχομαι σε ένα θεμελιώδες ε, ερώτημα του συναδέλφου Ντομινίκ Κρικέ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του ΣΑΝΤΟ, όπου έγιναν ορισμένες ε, ε, όπου συγκεκριμενοποιήθηκαν ορισμένα πράγματα, ε, πρέπει να ρωτήσουμε πώς, πώς γίνεται ο σχεδιασμός. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο προπολογισμού, όπως είπατε κι εσείς, αν υπάρξουν νέα εργαλεία, τι κάνουμε, αν ζητάμε από την Τράπεζα Επενδύσεων να μας βοηθήσει, τι κάνουμε λοιπόν. Επομένως, έχουμε το χρόνο με ένα διάλογο να δημιουργήσουμε αυτό το νέο ταμείο. Ε, αυτή η έκθεση θα είναι φιλόδοξη, αλλά θα σταθεί και στο ύψος των περιστάσεων και θα αποτελέσει απάντηση σε όλους αυτούς που τρίβουν τα χέρια ε, και υποστηρίζουν το Brexit είναι καλό πράγμα και θέλουν να δείξουν ότι η Ευρώπη είναι, θέλουμε να δείξουμε ότι η Ευρώπη είναι η απάντηση. Η Επιτροπή ε, των, μεταφορών δίνει απαντήσεις σε όσους ανησυχούν για τις περιφέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Η, η έκθεση είναι ανοιχτή σε τροποποιητικές προτάσεις μέχρι, το, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι. Δεν σας μένει πολύ καιρός, από ό,τι καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε και περνάμε αμέσως στις ε, κοινές, στους κοινούς κανονισμούς Κυρία Ντεμοντέ, ο, ο λόγος ε, είναι σε εσά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για μια έκθεση ανάλογη με αυτήν που μόλις συζητήσαμε. Και εδώ έχουμε μια επιταχυμένη διαδικασία και έλεγα ότι είναι ανάλογη η κατάσταση γιατί αφορά πάλι το Brexit και είναι γνωστό ότι το Brexit, ε, ε, ότι μάλλον η Μεγάλη Βρετανία επιθυμεί να εξέλθει της Ένωσης ε, τέλος Μαρτίου 2019 θα πράψουν να ισχύουν οι Ευρωπαϊκέ ρυθμίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό ισχύει και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Πρόκειται λοιπόν για έναν τομέα που ενδιαφέρεται πολύ και που εδώ πρόκειται για την αναγνώριση σε επίπεδο Ένωση των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες επιθεώρησης και ε, κάνουν ε, επισκέψεις ελέγχου στα πλοία που φέρουν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για αναγνωρισμένους οργανισμούς, τους οποίους κάθε δύο χρόνια επικυρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το εκάστοτε κράτος μέλος, που έχει ε, υποβάλει την αρχική αίτηση αναγνώρισης και καλείται χορηγός για να συνεχίσουν να διεξάγουν αυτές ε, τις επιθεωρήσεις. Αυτοί οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί θα πρέπει τουλάχιστον κάθε διετία να υπόκειται σε μια αξιολόγηση. Όμως το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον εξέλθει, δεν θα μπορεί πλέον να είναι χορηγός. Ε, αυτοί οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί δίνουν, ε, μάλλον λειτουργούν με βάση ε, συμφωνίες αναγνώρισης για όλες τις χώρες της Ένωσης. Άρα λοιπόν όταν εξέλθει το, Ευρωπα... το Βρετανικό η Βρετανία μάλλον, δεν θα μπορούν να προτείνουν ε, αναγνωρισμένους οργανισμούς για τα σκάφη που φέρουν τη δική τους ε, σημαία. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε αυτό το νομοθετικό κενό και η πρόταση της Κομισιόν είναι να τροποποιηθεί είναι η παράγραφος 8, ε, εδάφιο 1, Πρόκειται για τον κανονισμό 391 του 2009 και πρόκειται για την αντικατάσταση του κράτους χορηγού από, έναν, από τα κράτη-μέλη που έχει εγκρίνει και εξουσιοδοτήσει έναν από αυτούς τους αναγνωρισμένους οργανισμούς. Στην πράξη δηλαδή σημαίνει για κάποια, εγ, κάποιο είδους έγκριση ο κάθε, κάποιο κράτος μπορεί, οποιοδήποτε μάλλον κράτος μέλος μπορεί να θεωρηθεί ως ο χορηγός, ο εγγυητής ας πούμε αυτόν των εκάστοτε οργανισμών. Θα πρέπει λοιπόν να καλυφθεί αυτή, αυτό το νομοθετικό κενό που θα δημιουργηθεί με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι σημαντικό να διατηρηθεί η συνέχεια και προσθέτω και εγώ ε, ότι πρέπει να διατηρηθεί η συνέχεια και η λογική και η, δυνατό, η διαλειτουργικότητα για τους εφοπλιστές που ενδιαφέρονται. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια επιταχυμένη διαδικασία και γι' αυτό το λόγο επίσης η πρότασή μου είναι αυτή να εγκρίνουμε δηλαδή την αλλαγή χωρίς ε, τροπολογίες. Ελπίζω δηλαδή ότι θα είναι λιγότερο επίμαχη η κατάσταση από την έκθεση που μόλις εξετάσαμε, αλλά όπως σας είπα, βασική απέτηση είναι να προχωρήσουμε γρήγορα, ώστε να αλλάξει η νομοθεσία και να διασφαλιστεί η συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ντελμόντε. Κύριε Βαντεκάμπ, θέλετε το λόγο. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έχω την τιμή να μιλάω εκ μέρου του συναδέλφου Στέφαν Γκέρολτ που πρόσφατα εισήλθε στο Κοινοβούλιο για την επιθεώρηση πλέον όσον αφορά την αποχώρηση του Ινωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διατήρηση υψηλών προτύπων ασφαλείας είναι μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιθεώρηση και οι οργανισμοί επιθεώρησης δεν αποτελούν εξαίρεση. Όπως είπε η αγαπητή συναδελφό Ιζαμπέλ Ντεμόντι, υποστηρίζω την πρόταση της Επιτροπής χωρίς την πρόθεση να προτείνω τροπολογίε. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω τα εξής. Μετά από έρευνα του συστήματος του τελευταίου μήνες του συστήματος επιθεώρησης ε, των πλεόν και των επιχορηγήσεων υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ε, ε, κόστους και αποδοτικότητας. Υπάρχει επικάλυψη ευθυνών στην οδηγία ως προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών και την ε, παρακολούθηση, εποπτεία των οργανισμών επιθεώρησης, των αρχών επιθεώρησης. Είναι μια ε, δραστηριότητα την οποία ε, έχει αναλάβει ήδη η Επιτροπή και θα πρέπει η Επιτροπή να αποφασίσει αν θα απαλλάξει τα κρατημέλη από αυτή την υποχρέωση Επιπλέον, θα ήθελα από την πλευρά της Επιτροπής μια επανεξολόγηση της ε, χρηματοδότηση των κρατών μελών και θα πρέπει αυτό να απασχολήσει το Κοινοβούλιο στην έτου θητεία που θα ξεκινήσει το 2019. Η Επιτροπή θα ε, πρέπει να αξιολογήσει αν είναι πιο αποδοτικό οικονομικά οι οργανισμοί ε, συμβάλλονται άμεσα με την Επιτροπή χωρίς ε, να χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη. Αποκλεί τον ανταγωνισμό το χρηματοδοτικό μοντέλο μεταξύ των οργανισμών αυτών. Τώρα βλέπουμε την ανασφάλεια ως προς τις ευθύνες εξαιτίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως ένα κίνητρο για να, ένα κίνητρο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Τα μέτρα που προτείνονται αποτελούν ένα βήμα μπροστά για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που θα είναι επωφελής για όλους όσους συνεισφέρουν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον συνάδελφό μου Στέφαν Γκέρολ εκ μέρους του μάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντως είναι πολύ ταιριαστό γιατί έχουμε την ίδια κατεύθυνση και στις δύο εκθέσεις. Η Ζαμπέλα, ξέρω ότι είπε ότι θα πρέπει να μην προτείνουμε τροπολογίες για, αυτό, για αυτή την πρόταση. Όπως είπε και ο Βιμ, φαίνεται ότι θα, προτείνουμε, ή θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία, τη διαδικασία με συγχωρείτε, στο Συμβούλιο με μια πρόταση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αναφερθήκατε στην οδηγία 2015. Θα πρέπει να τις ε, επανεξετάσουμε είτε από την Επιτροπή είτε από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι διπλή δουλειά και εφόσον συζητήσουμε μια πρόταση τροπολογία στο Συμβούλιο, αυτό ήταν κάτι καλύτερο. Ίσως μπορούμε εμείς ως Κοινοβούλιο να προτείνουμε μια καλύτερα διατυπωμένη νομοθετικά πρόταση, ώστε να μπορούμε ταυτόχρονα να επανεξετάσουμε το θέμα. Και είναι σαφές ότι μπορεί να έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με μια πρόταση τροπολογίας, Δεν πρέπει απλά να το περάσουμε γρήγορα τα θέμα. Ε, Ενδεχομένω δεν είναι αμφιλεγόμενη αυτή η άποψη. Το ερώτημα είναι όμως ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής για αυτό το... και επίσης και η ίδια η, η συγγητρία Ισαμπέλα. Ευχαριστώ κυρία Μέισνερ. Η κυρία Σελιέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα στο όνομα της DG Move. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγήτρια για την γνωμοδότηση που αποτυπώνει τις φιλοδοξίες αυτής της πρότασης που αφορά τη νομική ανασφάλεια στην ε, επιθόρηση των πλοίων. Αυτή η πρόταση, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, θα πρέπει να εγκριθεί ταχύτατα. Είναι σημαντικό να επιλύσουμε την νομική αυτή ε, ανασφάλεια σύντομα. Και αυτή η πρόταση επίσης ε, συμπεριλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη τα οποία συνεργάζονται με τους σχετικούς οργανισμούς και που συμμετέχουν στην αξιολόγηση από την πλευρά της Επιτροπής της επίδοσής τους. Θα ήθελα να απαντήσω σε, σε αυτό που πρότεινε ο κ. Βαντελκάμπ και την παρέμβαση της κυρίας Μάισνερ. Σημειώνουμε την έκκλησή σας για την ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα και για τη δημιουργία ενός συστήματος γενικής εποπτείας. Οπότε, Λαμβάνουμε υπόψη τις προτάσεις και ανυπομονούμε παράλληλα σε σχέση με αυτή την πρόταση να ολοκληρώσουμε τις ε, διαβουλεύσεις. Η προτεραιότητα για εμάς είναι να ολοκληρώσουμε τις ε, συζητήσεις σε αυτό το, το φάκελο, αλλά παράλληλα λαμβάνουμε υπόψη και σημειώνουμε την ε, έκκληση για αύξηση της αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τελμόντα, έχετε το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις προτάσεις. Ε, Βέβαια θα πρέπει να συνδυάσουμε τις δύο απαιτήσει, δηλαδή η ταχύτητα, αλλά και εφόσον υπάρχει αυτή η έκκληση για περισσότερη αποτελεσματικότητα και μπορεί να λυθεί σε έφθετο χρόνο και απλά, νομίζω πως μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτήν, αυτή την οδό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να θυμίσω, ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 10 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Συνεχίζουμε. Όσον αφορά την απαλλαγή 2017 για την Επιτροπή και το σύνολο των οργανισμών και θα δώσω το λόγο στον κύριο Βιμ Βαντερκάμπ εξ ονόματος του κυρίου Προύστ και εξ ονόματος της Επιτροπής και στον κύριο Λεοντίνη για το σύνολο των οργανισμών. Και στη συνέχεια θα έχουμε μια συζήτηση μαζί σας με τους σκιώδεις εισηγητές και θα ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Βίμπαντεκάμπ, εσείς έχετε το λόγο πρώτα. Αγαπητοί συναδέλφοι, θα ήθελα να σας συγγνώμη για την απουσία μου και θα παρακαλώ στον Βήμα να διαβάσει αυτή τη δηλώση εκ μέρου μου. Υπέροχα. Η απαλλαγή για το, το, από τον προπολογισμό του 2017 είναι τεχνικό θέμα, επομένως ε, θα δώσω περιληπτικά ορισμένα ε, σημεία που νομίζω ότι αξίζει να ακούσετε. Καταρχάς, θα ήθελα να καλωσορίσω την ε, ενοποιημένη κατάσταση της Ένωσης, ακόμα και αν το το επίπεδο λάθους 2,4 ε, είναι πάνω από το επίπεδο του 2%. Ειδικότερα όσον αφορά στα ε, ζητήματα των μεταφορών. Θέλω να εκφράσω τη δυσαρέσκεια και τη λύπη μου ότι για τον τομέα της ανταγωνιστικότητας, ε, ανάπτυξης και απασχόλησης που είναι που ανήκει στον ε, στις μεταφορές. Το, το, το, το, Ελεκτικό Συμβούλιο δεν δίνει α, ε, περισσότερες πληροφορίες. Χαιρετίζω τα 9,3 ε, εκατομμύρια σε δεσμεύσεις και 3 εκατομμύρια σε πληρωμές που έχουν δοθεί το 2017. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή έχει επιλέξει 152 προγράμματα για να λάβουν χρηματοδότηση 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που αποδεικνύει την επιτυχία του προγράμματος. Εν κατεκλείδη, τα διάφορα ε, έγγραφα που μελετήθηκαν για την ε, ολοκλήρωση της ε, έκθεσης με κάνουν να σκεφτώ τα δύο πράγματα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Ο εσωτερικός έλεγχος της Επιτροπής ε, βρήκε αρκετές αδυναμίες στο, στο υπάρχον ζήτημα ε, ελέγχου της DigiMove για, τις, ε, για, την, για την αεροπορία και για τις μεταφορές. Έγιναν συστάσεις και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Και το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι η DigiMove αντιμετωπίζει δυσκολίες ε, στην πρόσληψη ε, εξειδικευμένων ανθρώπων οι οποίοι χρειάζονται για, να, για την ε, εξασφάλιση ενός ψηλού επίπεδου τεχνογνωσίας και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το παρακολουθούμε στενά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαντεκόμπ, ο κύριος Λοντίνη. Grazie Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή μας ε, καλείται να δώσει τη γνωμοδότησή της ε, προς την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού όσον αφορά την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για τη χρήση 2017. Τα σχέδια γνωμοδότησης που εγώ υποβάλλω σε εσά σήμερα αφορούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιας Ασφάλειας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αέρας, Ασφάλειας της Αεροπλοείας, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων, την Κοινή Επιχείρηση για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, το ΣΕΖΑΡ και την Κοινή Επιχείρηση Shift to Rail. Στη διάρκεια των ετών η διαδικασία απαλλαγή έχει, έχει καταστεί όλο ένα και πιο σημαντικό όργανο μέσο για να επαληθεύεται ο τρόπος με τον οποίο έχουν δαπανηθεί ε, τα δημόσια κονδύλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ελέγχει την εκτέλεση του προπολογισμού ε, των ευρωπαϊκών οργανισμών. Γίνεται λοιπόν έλεγχος των αιτήσεων ε, ομαδοποιημένων λόγω λογαριασμών της Ένωσης για την ετήσια έκθεση του, με βάση μάλλον την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση το, ε, τη δήλωση αξιοπιστίας. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι οι τρεις οργανισμοί και οι δύο κοινέ επιχειρήσεις ε, που περιλαμβάνονται σε αυτές τις νομοδοτήσεις έχουν διαχειριστεί τον προπολογισμό τους το 2017 με θεμητό και ε, κανονικό ε, τακτικό τρόπο. Μπαίνοντα τώρα στην ουσία των νομοδοτήσεων, η κοινή επιχείρηση Shift to Rail έφτασε σε ένα ποσοστό εκτέλεσης το 94% για τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων και 75% της υποχρεώσεις της επιστώσεις πληρωμών. Ε, ασχολείται με σύγκρουση συμφερόντων στα μέλη, στο προσωπικό του και στο αποσπασμένο του προσωπικό, καθώς επίσης και για τα μέλη του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εφαρμόσει μια στρατηγική κατά των απατών ad hoc που ενσωματώνει την ε, στρατηγική ορίζοντας 2020. Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την στην ασφάλεια της ναυτιλίας, την ασφάλεια στη θάλασσα, προτείνω να δεχτούμε θετικά τη σχέση ανάμεσα ε, στη Frontex και την Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον έλεγχο της αλληλείας που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2017 για να ε, ε, ελέγξει την αποτελεσματικότητα και τον τρόπο λειτουργίας των δύο οργανισμών 63,3 δις και στη διάθεσή της και 55,1 ε, δις πιστώσεις πληρωμών αντίστοιχο στο 97,32% του συνολικού προπολογισμού. Το 2017 δεν σημειώθηκαν ε, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας έχει προσεγγίσει την πλήρη εκτέλεση του προπολογισμού της με 99% ποσοστό εκτέλεση. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ότι στις δημόσιους διαγωνισμούς που σχετίζονται κυρίως με υπηρεσίες εντοπίστηκαν ελλείψεις που θέτουν σε κίνδυνο την σχέση ποιότητας τιμής. Επιπλέον υπογραμμίζουμε ότι η αναθεώρηση του βασικού κανονισμού του οργανισμού δεν άρχισε να ισχύει το 2017 όπως αρχικά είχε προβληθεί. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Σιδηρόδρομους έχει ε, φτάσει στο 100% εκτέλεσης για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και 93,3% ε, για τις πιστώσεις πληρωμών. Ο οργανισμός αυτός το είχε μάλλον πρόθεση να τροποποιήσει το δομή του για να εκτελέσει νέες αρμοδιότητες που ανατέθηκαν από το νέο πακέτο για τους σιδηροδρόμους και για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη στρατηγική κατά των απατών. Η κοινή επιχείρηση τώρα τέλος για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό Σέζαρ έφτασε 113 δις πιστώσεις υποχρεώσεων και 191 δις πιστώσεις πληρωμών. Ε, τα ποσοστά εκτέλεσης ήταν 80% και 69%. Ο χαμηλός, το χαμηλό ποσοστό γενικής εκτέλεσης οφείλεται βασικά σε καθυστερήσεις ή στην ατελή τιμολόγηση από πλευράς των ε, ε, βιομηχανιών για να μπορέσουν να μπουν εντός του ελαχίστου ορίου της δαπάνες, στις δαπάνες ε, λειτουργίας. Προτείνω λοιπόν να δοθεί η απαλλαγή για την εκτέλεση προπολογισμού για τη χρήση 2017 σε όλους τους οργανισμούς και στους ε, Εκείνε επιχειρήσει που περιλαμβάνουν οι δικέ μου γνωμοδοτήσει. 13 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Πρόεδρε και συνάδελφοι, σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και παραμένω στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεοντίνη. Κυρία Μάισνερ, θέλατε το λόγο. Μάλιστα. Δεν μπορεί να είναι εδώ ο κύριο και μου ζήτησε να διαβάσω κάποια σχόλια εκ μέρου του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγητές για το έργο τους και να ξεκινήσει με μια γενική παρατήρηση ότι στον τομέα των μεταφορών η έκθεση δείχνει μια καλή διαχείριση του ε, προϋπολογισμού και από την πλευρά τη και από του οργανισμούς. Υπάρχει περιθώριο ε, βελτίωσης, όμως το επίπεδο λαθών τίνει να μειώνεται και φαίνεται ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε καλό δρόμο. Αυτό φυσικά είναι κάτι πολύ θετικό και που θα πρέπει να, θα πρέπει να μας ικανοποιεί. Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα είναι καθαρά ε, δημοσιονομικής φύσης και δεν θα πρέπει να ε, μην, να μας αποτρέπει το να ε, δίνουμε έμφαση στην ουσία και στο του προπολογισμού. Παρακαλώ για ησυχία η ομιλήτρια. Όσον αφορά αυτό υπήρξαν ειδικέ εκθέσεις για τα δικαιώματα των ε, επιβατών, για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και θα πρέπει να τα αναλογιστούμε όλα αυτά όταν θα αξιολογήσουμε το, τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αν δεν το πράξουμε δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι. Η Επιτροπή και τα εκτελεστικοί οργανισμοί και ο σχόλιο στην πρόταση του κυρίου Προύστ θεωρεί ότι η επαναξιολόγηση του ε, μηχανισμού συνδέοντα στην Ευρώπη είναι κάτι που, θα, είναι σημαντικό γιατί υπάρχει χαμηλή, χαμηλό, ποσοστό ε, του προπολογισμού και πολλά γίνονται εκ μέρου του ΕΦΣΥ και όχι από την διευκόλυνση τη στην Ευρώπη. Όσον αφορά του οργανισμού και την γνωμοδότηση του κυρίου Λεοντίνη. Ο κύριο Τέλτσκα μπορεί να τα στηρίξει σε μεγάλο βαθμό και θα προτείνει μερικέ μόνο τροπολογίε ε, ε, που θα είναι σύμφωνα με τις γενικέ παρατηρήσεις του. Σα ευχαριστώ πολύ για την ώρα. Δεν έχουμε κανέναν από πλευρά τη Επιτροπή για να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα των απαλλαγών. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ε, ορίζεται στι 13 ε, Δεκεμβρίου στι 11. Κύριε Λεοντίνη, θέλετε να κάνετε κάποιες άλλες διευκρινήσεις, παρακαλώ. Μάλιστα. Σημειώνω θετικά τα όσα υπογράμμισε η κυρία Μέσνερ και εγώ τίνω να θεωρήσω πιο σκόπιμη μία πιο ποιοτική αξιολόγηση και λιγότερο αποκλειστικός οικονομικού τύπου ε, που βασίζεται λιγότερο στη σχέση ανάμεσα στην απόδοση και στο κόστος. Αλλά με τα στοιχεία που έχουμε, μόνο τέτοιου είδους εκθέσεις μπορούμε να κάνουμε και είμαι υπέρ της έγκρισης. Και ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα διακόψουμε για 15 λεπτά τώρα και στη συνέχεια θα έχουμε τους εμπειρογνώμονές μας που θα μας παρουσιάσουν την μελέτη για το Brexit, συνέπειες στον τουρισμό και τις μεταφορές και βεβαίως το σενάριο απουσία συμφωνίας. Ποιες θα είναι οι πραγματικές συνέπειες. Σας καλώ λοιπόν στις, σε 15 λεπτά να επανέλθετε και εντωμεταξύ να φροντίσουμε ώστε όλοι να μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτή την έκθεση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινούμε εκ νέου τη συνεδρίαση και ε, ξεκινάμε με την παρουσίαση της μελέτης από το, από το θεματικό τμήμα όσον αφορά το Brexit, ε, οι συνέπειες της περίπτωσης μη επίτευξης συμφωνίας, κυρίως για τον τομέα των μεταφορών αλλά και του τουρισμού. Αυτή η παρουσίαση συνεχίζει την ε, ακρόαση για, την, για τον αντίκτυπο του Brexit ε, και την περιμένουν διάφοροι εκπρόσωποι ε, του τομέα των μεταφορών που τους ακούσαμε το 2017 και το 2018 στην Επιτροπή μας. Τώρα, έχουν, εφόσον, επειδή υπάρχει λοιπόν συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, ε, γνωρίζουμε λοιπόν το κείμενο και, ε, και τον αντίκτυπο, ωστόσο περιμένουμε την απόφαση του Βρετανικού Κοινοβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου, ε, που αυτή τη στιγμή δεν είναι και το πιο προφανές πράγμα, Επομένω, δίνω το λόγο στους επιρρογνώμονες για να δούμε τι, τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση μη επιτεύξη συμφωνίας. Καλό λοιπόν τους, ε, ε, τους ανθρώπους που εκπώνησαν ε, την μελέτη αυτή, ο, ο κύριος ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα, ο κύριος Ραφαέλ Αλφόνσο, σας ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας εδώ και ο κύριος Μικέλ Τρονκόνσο Θερέρ, σας καλώ λοιπόν να μας παρουσιάσετε αυτή τη μελέτη. Θα σας δώσω το λόγο θα έχετε πέντε λεπτά και μετά θα ξεκινήσω την συζήτηση. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο, το λόγο στον κύριο Παπί, Παπί Φεράντο. Ε, θα ήθελα να ε, μιλήσω στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω τα βασικά συμπεράσματα της ε, μελέτης που κάναμε τους τελευταίους μήνες. Έχετε ένα αντίγραφο τη έκθεση στα χέρια σας, φαντάζομαι. Είναι μια μεγάλη έκθεση, 170 σελίδες, είναι αρκετά εκτενής. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε τις βασικές κατευθυντηρίες γραμμές ε, της μεθοδολογίας μας για την έρευνα και οι βασικές συστάσεις ε, που θέλουμε να ε, προτείνουμε σε αυτή την επιτροπή. Πρώτη διαφάνεια. Τρία τμήματα θα έχει παρουσίαση. Βλέπετε στις οθόνε σα. Το πρώτο στοιχείο στο οποίο θέλουμε να αναφερθούμε είναι η σημασία των οικονομικών σχέσεων μεταξύ του Μένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία της οικονομίας του Μεν Βασιλείου. Μιλάμε για μια, χρόνια που, χώρα που ε, έχει το 3% του ΑΕΠ. Έχουμε έλλειμμα στο εμπορικό συζύγιο του Ηνωμένου Βασιλείου ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση 110 εκατομμύρια ευρώ που είναι το 5% του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου και προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικός εταίρος του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την εμπορία αγαθών και ε, υπηρεσιών. Οι επενδύσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 48% ε, στο σύνολο 40% των επενδύσεων των Βασιλείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, βλέπουμε την ε, μεγάλη εξάρτηση μεταξύ των δύο οικονομιών και ειδικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με τις μεταφορές, τον τουρισμό και τον ταχυδρομικό τομέα που ε, είναι οι τρεις τομείς που καλύφθηκαν από την μελέτη μας. Ευχαριστώ πολύ. Στην οθόνη βλέπετε τώρα ένα γράφημα που δείχνει την εμπορία αγαθών μεταξύ των δύο γεωγραφικών περιοχών, ε, την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, έχουμε αφαιρέσει το Ενωμένο Βασιλείο. Βλέπετε, έχουμε μια σταθεροποίηση στο 50%. Επόμενη διαφάνεια. Όσον αφορά τη μεταφορά εμπορί, εμπορευμάτων, παρά τι επενδύσει και τη σημασία του, της ρίκας της μάχης, τα περισσότερα εμπορεύματα ε, μεταφέρονται από θαλάσσεις. Αυτό είναι κάτι το, στο οποίο θέλω να πιστήσω την προσοχή σας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Όσον αφορά τη μεταφορά επιβατών, υπάρχει ε, μεγάλος αριθμός ταξιδιών στα 50 εκατομμύρια περίπου από κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου σε, άλλες, σε άλλους προορισμούς ε, της Ευρώπης των 27. 24 επισκέπτες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο από άλλες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό είναι ότι όσον αφορά τα άτομα, τους επιβάτες, οι αερομεταφορές είναι ο κυρίαρχος τρόπος μετακίνησης. Στα εμπορεύματα έχουμε Μεταφορέ από θαλάσσει. Όσον αφορά τους επιβάτες όμως ε, κυριαρχούν ε, οι αεροπορικέ μεταφορέ. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. 32 εκατομμύρια επισκέψεις ε, πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλλον πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου κατοίκων στην Ευρώπη των 27. Συνολική δαπάνη κοντά στα 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίση επισκέψεις προς τον Ηνωμένο Βασίλειο που κατοίκου της Ευρώπης των 27 Ε, μιλάμε για ένα ποσό δαπάνης ε, υποδέστριο των 5 ε, ε, δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα δώσω το λόγο τώρα, το λόγο στον συνάδελφό μου, τον Ραφαέλ Αλφόνζη, όσον αφορά τον αντίκτυπο μιας, ε, ενός Brexit χωρίς ε, συμφωνία. Χωρίς συμφωνία το Μήνο Βασίλειο θα ε, γίνει απλά μια τρίτη χώρα και αυτό θα σημαίνει ότι θα υπάρχει κόστος και για τις δύο πλευρές, όχι μόνο για τον Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Φυσικά το κόστος για την Ευρώπη των 27 στο σύνολό του θα είναι χαμηλότερο και δεν θα είναι αναλογικό με αυτό που θα πρέπει να υποστεί το Βασίλειο σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές αναφορές που έχουμε, μέχρι το 2030 οι σωρευτικές απώλειες σε ΑΕΠ θα είναι 0,44% για την Ευρώπη των 27% και 4,2% για το Ηνωμένο Βασίλειο αν λάβουμε υπόψη ένα απεσιόδοξο σενάριο. Όσον αφορά τον τομέα μεταφορά εμπορευμάτων, ε, μια μη συμφωνία θα προκαλέσει προφανώς κόστη που θα έχουν να κάνουν με δασμολόγηση και μη δασμολόγηση και ε, μια γενικότερη μείωση του όγκου των ε, εμπορευμάτων. Μεταφορές επιβατών και τουρισμός δύο τομείς που συνδέονται. Φυσικά θα είναι πολύ αρνητικός αντίκτυπος στη γενική μείωση, ε, στην ευκολία του ταξιδιού. Και πιο αρνητικά θα επηρεαστεί ο τομέας της, αερο, της πολιτικής αεροπορίας. Γιατί δεν υπάρχουν κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που να καλύπτουν αυτό το τομέα των αερομεταφορών. Πάμε στο νομικό ε, σκηνικό, να δούμε τι έχει γίνει σε θέματα νομοθεσίας. Βλέπουμε ότι στο μέτωπο μεταφορών ε, η τρέχουσα ε, νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χρειαστεί μεγάλε τροποποιήσει, γιατί δεν γίνεται ειδική αναφορά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμω είναι ένα περίεργο, περίπλοκο συμπέρασμα γιατί παρόλο που δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη εξορισμού, θα χρειαστούμε προσαρμογές, θα χρειαστούμε συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου. Και ένα παράδειγμα είναι είναι ο κανονισμός για τις αεροπορικές υπηρεσίες που έχει να κάνει με την ε, αγορά της πολιτικής αεροπορίας, θα χρειαστούμε μια νέα συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου και Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορούν οι αερομεταφορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργούν ελεύθερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι περίπλοκη κατάσταση. Επίση, εξαρτάται από το τι θα πράξει το Ηνωμένο Βασίλειο με τη δικιά του νομοθεσία, με την έννοια ότι αν ε, μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, η ευρωπαϊκή νομοθεσία και αυτή η νομοθεσία δεν ε, τροποποιηθεί ως συνέπεια του Brexit, θα συνεχίσουν να ισχύουν ε, οι κανόνες. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι θα συμβεί. Επόμενη διαφάνεια. γενικές επιπτώσεις ε, για τον ε, των μεταφορών όσον αφορά τους κανόνες του καμποτάζ δεν θα ισχύουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Βασίλειο και οι συνέπειες θα είναι η μείωση της διαλειτουργικότητας και η μείωση του ε, ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών, δεν θα διασφαλίζονται όταν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωση ταξιδεύουν, θα χρησιμοποιούν ε, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά το TNT δίκτυο, θα υπάρξουν φυσικά εμπόδια και καθυστερήσεις και μπορεί να προκύψουν πιο σοβαρά θέματα ε, σε σχέση με το... Ε, με τις έργα και το, στην τριτομική γραμμή του Μπέλφαστ. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και τη διευκόλυνση συνδέοντα ε, την Ευρώπη, αναμένεται να συνεχίσουν να παρέχουν στο μέλλον ε, κατάλληλη χρηματοδότηση για το δίκτυο. Όμω υπάρχει ανασφάλεια. Και όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες, τους οργανισμούς ε, που έχουν να κάνουν ε, με το μέτρο μεταφορών και στους οποίους συμμετέχει το Μένο Βασίλειο, θα συνεχίσουν να συμμετέχουν εφόσον επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων χωρών. Στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, εκεί θα έχουμε αντίκτυπο και στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό σε σχέση με λειτουργικά τμήματα του εναέριου χώρου. Θα έχουμε κατακαιρματισμό του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και λιγότερο αποτελεσματική διαχείριση του εναέριου χώρου. Σε γενικές γραμμές θα υπάρξουν ρυθμιστικοί περιορισμοί που θα περιορίσουν ε, το δυνατότητα επέκταση και ανάπτυξη των αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την δικτυσιακή δομή, το σενάριο της μη συμφωνίας θα δημιουργήσει πρόβλημα γιατί κάποιες ε, αεροπορικές εταιρείε με συγκεκριμένη ιδιοκτησιακή δομή θα έχουν προβλήματα γιατί θα πρέπει να προσαρμοστούν οι κανόνες. Περνάμε στην επόμενη διαφάνεια όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, την αυσιπλοεία και την ε, χώρια αυσιπλοεία δεν ε, αναμένεται να υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας στα λιμάνια του Ηνωμένου Βασιλείου εις βάρος των ευρωπαϊκών ε, λιμένων γιατί ήδη τα ε, λιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υποδιαχείριση ιδιωτικών φορέων η εφαρμογή των κανόνων του ΩΣΑ αποκλείουν αλλαγές σε σχέση με την πρόσβαση ε, των χωρών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την πρόσβασή τους στα, στους λιμάνες του Νομένου Βασιλείου. Οι φορείς του Νομένου Βασιλείου και τα καταχωρημένα σκάφη δεν θα έχουν το δικαίωμα πλέον να να λειτουργούν ε, στους, ε, στην εσωτερική ε, συμπλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία 9650 δεν θα ισχύει πλέον σε σχέση με τα πιστοποιητικά κυβερνήτη σκάφους. Θα τεθούν εκτός ισχύης. Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Ορισμός Ασφάλειας στην Ναυτιλία, η λειτουργία του, η λειτουργία της ΕΜΣΑ δεν θα αλλάξει δραστικά. Και σε σχέση με τη ΣΕΣΝΗ, την Επιτροπή για τη Δημιουργία Κοινών Προτύπων στην χώρια ναυσιπλοεία, θα μπορούσε να επιτρέψει το Μένο Βασίλειο να συμμετέχει ως κράτος παρατηρητής. σιδηροδρόμους. Αρνητική επίπτωση θα έχουμε στην αλυσίδα φοδιασμού επειδή νέες διαδικασίες και νέοι συνορικοί έλεγχοι θα πρέπει να εισάγουν νέες ε, διαδικασίες που θα δημιουργούν καθυστερήσεις. Και όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση του συνδρομικού διαδρόμου εμπορευμάτων, κανονισμός 913 του 2010, αυτός ο διάδρομος δεν θέλει υπό την διαχείριση αυτού του κανονισμού και φυσικά η εταιρεία Eurostar και άλλες εταιρείες που συνεργάζονται με το Eurotunnel, στην συνοριακή έλεγχη και η νομοθετική απόκληση θα τις επηρεάσουν αρνητικά ως προς την ανταγωνιστικότητά τους. Οδικές μεταφορές. Εκεί θα χρειαστούμε εναρμόνιση των διατάξεων για την πρόσβαση στην αγορά και την πρόσβαση στο επάγγελμα των οδικών μεταφορέων και αυτό είναι βασικό θεμελιώδες για να διασφαλίσουμε μια αδιάσπαστη παροχή υπηρεσιών. Οι κατευθύνες γραμμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν ε, έναν τρόπο να επιτευχθεί με τέτοια εναρμόνιση. Όσον αφορά τα πρότυπα εκπομπών για τα οχήματα, δεν αναμένεται δραστική αλλαγή ε, τους ε, κανόνες ε, για οδήγηση και χρόνους ανάπαυσης. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος προσανατολισμό αυτή τη στιγμή και επομένως δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ποια θα είναι η κατεύθυνση που θα πάρει το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με αυτό το θέμα. Τουρισμός. Σχετίζεται πολύ στενά με το τι θα συμβεί με τη μεταφορά με τη μετακίνηση των επιβατών. Θα υπάρξουν ε, διαδικασίες ε, που θα δυσχεραίνουν την κατάσταση όπως συνολική έλεγχη και τα λοιπά που θα αυξήσουν το κόστος του ταξιδιού και την ποιότητα των υπηρεσιών. Συνορική έλεγχη και διαδικασίες θα μειώσουν την ευκολία του ταξιδιού των τουριστών. Το δικαίωμα παραμονής δεν περιορίζεται μονάχα στον τουρισμό. Υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα ακόμα. Επόμενη διαφάνεια. Ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η κατάσταση μετά το Brexit θα ρυθμίζεται από τους κανόνες που έχουν υιοθετηθεί από την UPU και τον ΣΕΡΠ. Όμως υπάρχουν υποχρεώσεις που έχουν ε, που έχει αναλάβει το Βασίλειο στο πλαίσιο της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση σε αυτές. Επίσης το Μελ Βασίλειο ε, αποφάσισε να παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα για τη δημιουργία και την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και ο κανονισμός για την ιστορική παράδοση ε, δεμάτων δεν θα δεσμεύει πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμω αναμένεται αυτό ο κανονισμό να ε, μεταφερθεί, να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίση, αναμένεται το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ευθυγραμμίσουν τα τεχνικά πρότυπα στι ταχυδρομικέ μεταφορέ. Και τέλος, νέοι τελωνικοί έλεγχοι και διαδικασίες για τη συλλογή του ΦΠΑ σε διασυνοριακές ε, επιχειρήσεις θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ. Είναι δύσκολο να παρουσιάσουμε τα πάντα που έχει καλύψει αυτή η έκθεση. Σε το σύντομο χρόνο υπάρχει ένα σημείο που έχουμε καλύψει, το σημείο 11, όπου έχουμε 10 διαφορετικές ε, μελέτες για διαφορετικές χώρες. Έχουμε κάνει μια αξιολόγηση του αντικτύπου ενός τέτοιου σενάριου στις 10 χώρες. Προτείνω να περάσουμε όμως στις ε, βασικές συστάσεις και να κάνουμε μια σύνοψη για τα γενικά συμπεράσματα της μελέτης. Όσον αφορά τις αερομεταφορέ, έχουμε το πιο δύσκολο σημείο. Είναι σημαντικό να ε, ξεκινήσουν γρήγορα διαπραγματεύσει σε μια περίπτωση μη συμφωνία. Υπάρχει ανάγκη ταχύστατα να πετύχουμε κάποια συμφωνία ώστε το σύστημα και η ροή των αερομεταφορών να συνεχίσει απρόσκοπτα. Έχω τέσσερα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη. Αντικατοπτρίζουμε την τρέχουσα συμφωνία μια διμερή συμφωνία δηλαδή μεταξύ της Ευρώπης των 27 και του Βασιλείου, να μην υπάρχουν ε, διαταραχέ. Επίση αυτό θα περιλαμβάνει και την πρόσβαση σε τρίτε χώρε πρόσβαση από τρίτε χώρε. Αυτό όμω είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν εταιρείε που έχουν ε, μετόχου από διαφορετικέ ε, περιοχέ, Αυτό θα πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Όσον αφορά την ναυτιλία και τις περιπτώσεις του καμποτάζ, Υπάρχει επίγουσα ανάγκη για ταχύστατες, ε, τάχιστες συμφωνίες σε περίπτωση μη συμφωνίες τον συνδυαμικό τομέα. Ο συνάδελφός μου, ο κ. Αλφόνς, ήδη διερεύνησε πώς θα μπορούσε αυτό να προκαλέσει δυσκολίες στη σύραγγα της μάχης και χρειάζεται ε, επομένως και σε αυτό το τομέα μια γρήγορη συμφωνία δεν υπάρχουν μεγάλες ε, δυσκολίες στον οδικό κλάδο γιατί η νομοθεσία που εφαρμόζεται είναι συμφωνεί και με τη συμφωνία στο πλαίσιο του Οργανισμού Εθνών, στις οποίες συμμετέχει και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στον τουρισμό υπάρχει επίσης ανασφάλεια. Θα εξαρτηθεί από τις, ε, τα επόμενα βήματα. Αν θα θέλουν να κρατήσουν μια εύκολη πρόσβαση, γρήγορο έλεγχο, γρήγορες ουρές με την επίδειξη απλώς του διαβατηρίου. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε ε, να δούμε αν θα υπάρξουν ε, ε, περαιτέρω θεωρήσεις ε, ή έλεγχη. Αυτό ξερετε όμως πάντα από την ύπαρξη καλής διάθεσης από την πλευρά των δύο μερών την πρώτη μέρα της ε, ε, εξόδου χωρίς συμφωνία. Ταχυδρομικές ε, υπηρεσίε και εκεί χρειάζονται πάλι γρήγορε συμφωνίε γιατί αλλιώ δεν θα υπάρχει εγγύηση ότι ένα πακέτο θα φτάσει από εδώ στο Λίτς και ότι θα μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να δει πού βρίσκεται το δέμα και πότε θα παραδοθεί. Από όλα τα κράτη-μέλη, οι υπηρεσίες παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Χρειάζεται λοιπόν γρήγορη συμφωνία, το συντομότερο δυνατό. Ποιε θα είναι οι στάσεις που θα κάνουμε στην Επιτροπή σας και ίσως ε, ξεπερνάμε λίγο τα όρια και σας λέμε πολλά. Οι συστάσεις μας είναι να δημιουργηθεί ένα επικοδομητικό κλίμα γιατί υπάρχουν ε, αμοιβέ επιπτώσεις Άρα χρειάζεται ένα θετικό πνεύμα και αν υπάρχει κατανόηση και από τα δύο μέρη ότι έχει συμβεί κάτι άσχημο θα πρέπει να υπάρξει γρήγορη αντίδραση για να ε, διευκολυνθεί η κατάσταση. Αυτό το τονίσαμε και τη διάρκεια της παρουσίασης. Και από νομικής πλευράς Θα δώσω το λόγο στον αδελφό μου, γιατί ξέρει πολλά προστερά από εμένα, αλλά μια γρήγορη συμφωνία θα μπορούσε να γίνει μέσω διμερών συμφωνιών, κάτι που μπορεί να λάβει χώρα έχετε και αυτή είναι η δεύτερη σύστασή μας, να παρέχετε τη στήριξή σα σε αυτές τις διμερείς συμφωνίες σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη. ολοκληρώνοντα θέλω να σα ευχαριστώ για όλη την στήριξη που είχαμε από το θεματικό τμήμα. Ήταν πολύ μεγάλη βοήθειά σας. Τέσσερις ήμασταν συντάκτες. Είχαμε και πέντε εμπειρογνώμονες ε, που εξέτασαν την ε, έκθεσή μας. Σας, ενθαρρύνω να τη διαβάσετε και ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Merci Σας ευχαριστώ για αυτή σας την παρουσίαση που πραγματικά μας προκαλεί ρίγη και μας οδηγεί να πούμε ότι οι συνέπειες στον τομέα των μεταφορών θα είναι καταστροφικές. Αυτό είναι το συμπέρασμα αυτής της μελέτης. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και καταστροφικός αντίκτυπος δεν σταματά στον τομέα των οδικών μεταφορών ή στους σιδηροδρόμους, αλλά και στην αεροπλοεία επηρεάζει και τον, θα, τις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση θα προχωρήσουμε στη συζήτηση. Κύριε Πίπερ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Ήταν εντυπωσιακό αυτή η διασύνδεση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και τις υπόλοιπε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι όπως παρουσιάστηκε. Και ειδικά για το τομέα των μεταφορών και του τουρισμού θα είναι δραματικές οι επιπτώσεις όπως ε, μας το παρουσιάσατε. Θεωρώ όμως ότι, πρέπει, ότι έχουμε προχωρήσει λίγο παραπέρα, γιατί όταν ακούμε κάτι τέτοιο, το καλύτερο σε αυτό είναι να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, φυσικά, υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε σε μη συμφωνία, έξοδο χωρίς συμφωνία και το ερώτημά μου είναι κάτι που ακούγεται από πολλές ε, πλευρές και διάφορα υποτιθέμενα σενάρια. Στις αερομεταφορές θα υπάρχει μια διμερή συμφωνία και δεν θα είναι πρόβλημα αυτό να συμβεί. Οι αεροπορικές εταιρείε έχουν προσανατολιστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Η British Airways ε, κατά 50% ε, έχει δικτυθεί από άλλα κράτη-μέλη και από ό,τι καταλαβαίνω, ίσως το βλέπετε διαφορετικά εσείς, θα πρέπει να ασκηθεί πίση και η και άλλες εταιρείε να έχουν έτοιμα τα προγράμματα τους για τους επόμενους μήνες. Όσον αφορά τους ιδιοδρόμου και εκεί υπάρχουν σενάρια διμερείς συμφωνίες και εκεί υπάρχουν σχέδια σε περίπτωση αποτυχίας, εφεδρικά σχέδια. Αυτό που μου δημιουργεί ε, έκπληξη είναι οι οδικές μεταφορές όπου εκεί βλέπω εγώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί τα πολλά φορτηγά θα πρέπει να ελέγχονται σε περίπτωση μη συμφωνίας και αν κλείσει το αυτοκινητόδρομο στον Ντόβερ, τότε εκεί θα, έχουμε, θα βιώσουμε ένα τεράστιο δράμα σε περίπτωση μη συμφωνίας. Στους άλλους τομείς θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να βρούμε λύσεις. Αλλά αυτό που εύχομαι και αυτό που πιστεύω ότι πολλοί ακόμα εύχονται είναι να υπάρξει ένας τρόπος να κρατήσουμε τους Βρετανούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα αξιολογείτε αυτό εσείς με τα εφηδρικά σχέδια για τους διαφορετικούς τομείς μεταφοράς. Πώς είναι οι διαπραγματεύσεις Πώς θα μπορέσουμε από τη μία μέρα στην άλλη να εφαρμόσουμε τις νέες συμφωνίες. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποια είναι η εκτίμησή σας για τις οδικές μεταφορές. Ίσως και εκεί θα μπορούσατε να επιλογίσετε κάπως καλύτερα γιατί είναι, θεωρείτε ότι είναι εκεί το μικρότερο πρόβλημα Euh, Ευχαριστούμε κύριε Επίπερ. Η κυρία Δελμόντε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για αυτή την έκθεση και τα γραφήματα. Εγώ θέλω να επανέλθω στο θέμα του αντικτύπου ε, για τη στις μεταφορές για να γνωρίζω ακριβώ αν, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσατε. Είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις εισαγωγές, εξαγωγές. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που θα μπορούσαν να επηρεάσουν, όπω εξωτερικοί παράγοντε που θα μπορούσαν να αλλάξουν, να επηρεάσουν αυτά τα στοιχεία. Πέρα βέβαια από το γεγονό ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία. Και δεύτερον, κατά τη γνώμη σα υπάρχουν τομεί που θα ωφεληθούν εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Δεύτερη μου ερώτηση αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε ήδη ε, εξετάσει. Ε, δηλαδή, σύμφωνα με τα ε, συσχύουσες προδιαγραφές θα μπορούσε να ισχύσει η υπόθεση μιας μεταφοράς των Βρετανικών αεροπορικών εταιριών εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Έχετε αξιολογήσει και αυτό του είδους την υπόθεση και τι αντίκτυπο θα έχει αυτή. Και τρίτη ερώτηση αφορά μια ιδιαίτερη περίπτωση που πήρε μεγάλη δημοσιότητα στις εφημερίδες το είναι το θέμα του Γιβραλτάρ ε, όπου επικρατούν πολλές εντάσεις ανάμεσα στην Ισπανία και την Μεγάλη Βρετανία. Έχετε κάνει κάποια μελέτη εδώ, κάποια αξιολόγηση, ποια επίπτωση θα έχει αυτό στις συνθήκες εργασίας. Ήδη υπάρχουν δυσκολίες για τη μεταφορά ας πούμε, εργαζομένων που πρέπει να, αυτό το, να διασχίσουν αυτό το σύνορο το γεωγραφικό. Και αν υπάρχουν επίσης επιπτώσεις για, αυτού του, για, για τις ε, υπερπεριφερειακές περιοχές. Ποιες είναι οι δικές σας ε, σκέψεις λοιπόν για αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία ε, Ντελμόντε, κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν ε, μπορούσα να διαβάσω όλη την εξήγητη που υποχρεώσει. Μας το παρουσιάσετε πολύ αναλυτικά. Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν ε, οι αερομεταφορείς πρώτοι που ήρθαν σε επαφή μαζί μας που είπαν ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί ο τομέας αυτός, γιατί θα ήταν πραγματικά καταστροφικό. Είχαμε φυσικά και ακροάσεις για κάθε τομέα μεταφορών και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως είπε και ο κύριος Πίπερ. Δεν απορώ ότι υπάρχουν ήδη εφεδρικά σχέδια. Είναι απαραίτητο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στο θέμα των μεταφορών, ώστε να υποστηρίζουμε ένα remain και μπορεί να συμβεί, όμως δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Και στην περίπτωση μη συμφωνίας επίσης, θεωρώ ότι η έξοδο χωρί συμφωνία θα δημιουργήσει πολύ μεγάλε δυσκολίε και για τον Βασίλειο και για την Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να είμαστε προετοιμασμένοι. Και βασικά έχω δύο ερωτήσει είναι αυτό που είπε ο κύριος Πίπερ, τι θα γίνει με τα διάφορα ε, μπλοκαρίσματα που θα υπάρξουν στις οδικές μεταφορές, με τα φορτηγά. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά τις ε, νέες μεταφορές. Είπατε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολο η ΆΣΑ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο με τις πιστοποίησεις άλλων οδών, όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές. Συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των μεταφορών στην ομάδα αυτή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάισνερ. Ο κύριος Κοχ, έχετε εσείς το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις επεξηγήσεις και για την έκθεσή σας. Όλοι γνώριζαμε ότι και οι δύο πλευρές έχουν να, να χάσουν, ειδικά στην περίπτωση μη συμφωνίας. Τώρα γνωρίζουμε πολύ καλά τι θα συμβεί. Όμως, ο πληθυσμός δεν το γνωρίζει και θα διαβάσει όλες αυτές τις σελίδες. Τι θα κάνουν οι πολίτες με το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στον οδικό τομέα και στην Ευρώπη και στην Μεροβασίλεια. Ίσως υπάρξει ένα αποτέλεσμα ίσως θα πρέπει να μάλλον ρωτήσει η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας τους πολίτες αν το ήθελαν αυτό, αν το ήθελαν αυτό με όλε τι αρνητικέ συνέπειες. Πρέπει να το γνωρίζουμε εμεί, αλλά πρέπει να το γνωρίζει και το κοινό. Κύριε σας ευχαριστώ πολύ για την ε, έκθεση. Δεν, ε, άκουσα, ε, δεν την άκουσα όλη, ωστόσο θεωρώ ότι ελπίζουμε ότι οι συνέπειε σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία δεν θα είναι τόσο μεγάλε. Είναι κάτι όμω το οποίο πρέπει να ετοιμαστούμε και η Επιτροπή μάλιστα ε, προετοιμάζεται σε περίπτωση που τα πράγματα καταλήξουν εκεί. Όσες χώρες έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο ή σχέσεις ε, ή εξαρτώνται ε, ή έχουν σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατά κάποιο τρόπο προετοιμάζονται και νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επίση. Επομένω, ε, νομίζω υπάρχει μία απόκριση από όλα τα μέρη. Γνωρίζουμε ε, τα προβλήματα της αεροπορίας και των λιμανιών. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε έγγραφα όπως και αυτό, ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς ε, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση μη ύπαρξη συμφωνίας και τι αυτό θα τι, τι σημαίνει για τους α, ε, ε, Βρετανούς. Α, ψηφίσαν ορισμένα πράγματα, θα ψηφίσουν και άλλα την επόμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, λοιπόν, νομίζω ότι αυτό αυτή η μελέτη θα μας δώσει τις επαρκείς οδηγίες για το πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος τον κύριο Ρικέ. Ως προς το πρώτο σχόλιο, η υποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ε, θα γίνει ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Το δεύτερο σχόλιο είναι το εξής. Αν δεν είμαστε ικανοί να μάθουμε περισσότερα πράγματα σε χρόνο τριών ετών, για παράδειγμα, θα είναι πολύ πιο περίπλοκο να έχουμε διαπραγματεύσεις ε, μετά το πέρας αυτού του ε, χρονικού περιθωρίου. Τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα τότε. Όσον αφορά στις δεμερείς σχέσεις, νομίζω ότι ε, εάν πρόκειται για διμερείς σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ' εξαίρεση, ε, δεν νομίζω τα πράγματα θα, ε, έχουν γρήγορους, θα, θα γίνουν με γρήγορους ρυθμούς. Οι διμερείς σχέσεις δεν υπάρχουν στο, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι σε ό,τι, περνά από την Ευρωπαϊκή Ένωση την, αυτή καθευτεί υπάρχει μια κοινοβουλευτική επιτροπή ε, και υπάρχει μια συζήτηση και απαιτείται μια συζήτηση με, με, το, ε, με το νομοθετικό τρίγωνο Κοινοβουλίου, ε, Συμβουλίου και Επιτροπής και αυτό ε, έχει και τις δικές του δυσκολίες. Επομένως, οι διμερείς σχέσεις δεν, ε, οι διμερείς συμφωνίες, συγγνώμη, δεν ε, είναι επιτυχείς. Γιατί αυτές θα πρέπει επίσης να ψηφιστούν. Προσωπικά, ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμο, γιατί θα ήταν καταστροφικό ε, ε, κάτι τέτοιο. Ε, θα ήθελα να πω τελειώνοντας, ότι ό,τι δεν καταφέραμε να κάνουμε σε τρία χρόνια, δεν νομίζω ότι το καταφέρουμε σε τρεις μήνες. Τώρα το λόγο κύριο Στέμπορκ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ολοκληρωμένη μελέτη ε, με σαφείς ε, προτάσεις. Έχω ωστόσο μία ερώτηση ε, στον τομέα της ε, αεροπορίας. Σε περίπτωση λοιπόν μη συμφωνίας, οι ε, αεροπορικές εταιρείε του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ένα πλεονέκτημα το οποίο θα είναι άδικο, μπορούσαμε να πούμε. Νομίζω το ίδιο μπορεί να, να πούμε και για, για τους υπόλοιπους τρόπους μεταφοράς. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις για εκείνο το κατά κάποιο τρόπο άδικο πλεονέκτημα ε, τι σημαίνει αυτό, πώς θα μπορούσαμε να, ε, ανταγωνιστούμε τις ε, αεροπορικές εταιρείε του Ηνωμένου Βασιλείου, πώς αυτό θα επηρεάσει τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εταιρείε. Και επίσης, αν έχει γίνει αξιολόγηση, ποια είναι τα συμπεράσματά σας γιατί αυτό νομίζω αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την Ευρώπη των 27. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις που θέλετε να θέσετε. Όχι, εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Θα μπορούσατε να μας πείτε με σαφήνεια ποιες θα είναι οι περιοχές που θα, ε, στις οποίες θα υπάρχει άμεση, άμεσος αντίκτυπος το πρώτο τα πρώτα σύνορα είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο, κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι στη Γαλλία. Άρα ποιε θα είναι οι περιοχές που θα υποστούν τις συνέπειες και αναφορικά τώρα στους τομείς. Γιατί εδώ υπάρχουν κάποια, κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ε, στην Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες συνέπειες που δεν θα υπάρχουν σε άλλες περιοχές. Επομένως, θα θέλουμε να μας πείτε τις συνέπειες σε περιφερειακό επίπεδο. Το δεύτερο ερώτημα, συνεχίζοντας το, τις παρεμβάσεις του κ. Πικέ και του κ. Ρικέρ, αν υπάρχουν λοιπόν διμερείς ε, συμφωνίες, τότε εδώ έχουμε πρόβλημα... Yes. Not... Έχουμε πρόβλημα χρηματοδότησης, διότι ε, δεν σχετίζεται το Κοινοβούλιο θα ήθελα λοιπόν ε, ε, ε, να σας πω ότι όσον αφορά στη δική μας επιτροπή αυτό θα, θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα. Το τρίτο ερώτημα είναι το εξής. Μπορούμε να έχουμε γνώση σήμερα του πόσο μπορεί να μας κοστίσει όσον αφορά στον τομέα των υποδομών ε, για να υπάρξει καινούριο, να υπάρχουν καινούργια σύνορα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Πώς θα γίνει, ε, πόσο θα κοστίσει κάτι τέτοιο. Και θα σας αφήσω να μας δώσετε τις απαντήσεις. Ε, ο κύριος Παπί έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολλά τα ερωτήματα, ελπίζω να μην ξεχάσω κάποια από αυτά. Θα ξεκινήσω από το πρώτο και καλό λοιπόν και τους συναδέλφους μου να, να, να, εκφράσουν ότι, ότι θέλουν εκείνοι να σχολιάσουν. Ε, στους ε, συναδέλφους λοιπόν, όταν είπαμε ότι είναι λιγότερο δύσκολο σε περίπτωση του, τομέα, τον, ε, του δικού τομέα, ε, είναι ότι σε σχέση με του άλλου τομεί χρειαζόμαστε μια νομική βάση. Ενώ στο νομικό τομέα, στον οδικό τομέα υπάρχει ήδη μια νομική βάση. Ε, εάν δεν θέλετε να σταματήσετε στα σύνορα, δεν τα σταματάτε. Αν θέλετε να έχετε ένα ελαφρύτερο εντό εισαγωγικών ε, σύνορο, τότε μπορείτε να το έχετε μέσω τυχαίου ελέγχου, μέσω δειγματοληπτικού ελέγχου. Ενώ το πρόβλημα για του άλλου τομεί είναι ότι χρειαζόμαστε χαρτί, χρειαζόμαστε νομοθεσία. Έχουμε, θα χρειαζόμαστε επισήμω ε, εγκεκριμένα έγγραφα, κάποια νομική βάση. Επομένως, γι' αυτό νομίζουμε ότι στους άλλους τρεις τομείς ε, υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με τον ε, οδικό τομέα. Αναφορικά τώρα με τους ε, αριθμούς, ε, το είπαν και συνάδελφοί σας χρησιμοποίησαμε εργαλεία που ήταν διαθέσιμα από τη Eurostat, γιατί δεν είχαμε ε, στο πλαίσιο των τεσσάρων μηνών να ξεκινήσουμε μια οικονομική συλλογή δεδομένων. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο αυτό. Αλλά υπάρχουν επαρκή δεδομένα από το Eurostat στη διάθεσή μας, τα οποία χρησιμοποίησαμε και δευτε, δευτερευόντως υπάρχει μια έκθεση από τον ε, καθηγητή Μπέλγκεν στο ε, Ινστιτούτο του Έσεν το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη βιβλιογραφία. Και αυτή η έκθεση μάλιστα έχει κάνει τις, ε, τις πιο... Ε, τις καλύτερες ε, εκτιμήσεις για το, τον αντίκτυπο στον ΑΕΠ ότι ενδεχομένως στην Ευρώπη των 27 ίσως υπάρχει μία μείωση της τάξης 0,4 ενώ ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο ίσως υπάρχει μία μείωση του 4, βαθμών ε, ε, στο ΕΕΠ, στη μονομιάς. Εάν λοιπόν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, ε, μπορείτε να τις βρείτε στη βιβλιογραφία. Δεν προχωρήσαμε σε αναλυτική κατάσταση του, ε, της, της, κατάστασης με το, με το Γιβραρτάρ, γιατί σε εκείνο το στάδιο ε, είχαν κλείσει οι διαπραγματεύσεις και δεν υπήρχε ε, συμφωνία, επομένως δεν είχαμε το χρόνο να συμπεριλάβουμε κάτι τέτοιο. Ίσως ε, για τους επιμέρους τομείς μπορώ να σου δώσω το λόγο, Ραφαέλ, για να εξηγήσει πώς θα μπορούσαν οι τομείς πολιτικής αεροπορίας πώς θα μπορούσαν να αποφεληθεί από την μη ύπαρξη συμφωνίας. Θα μπορούσαν και αυτό μια περίπτωση, αλλά σε γενικέ γραμμέ δεν ε, περιμένουμε κάποια πλεονεκτήματα αναφορικά με αυτό σαν αφορά την αυτιλία και τον τομέα των αερομεταφορών θεωρούμε ότι σε γενικέ γραμμέ θα μπορούσε να υπάρξει μείωση στον ανταγωνισμό παντού και στο Βασίλειο και στην Ευρώπη των 27, γιατί θα έχουμε να κάνουμε με μια μικρότερη συγκεκριμένη αγορά, χαμηλότερο αριθμό εταιριών και ανταγωνιστών είναι σημαντικό να υπάρξει πολιτική βούληση για να δημιουργηθεί η νομοθετική βάση ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Χωρί την νομική βάση είμαστε με τα χέρια δεμένα. Εκτιμώ πολύ αυτό που είπε και παρουσίασε ο κύριος Ερικέ και πράγματι η νομοθετική διαδικασία χρειάζεται πολύ χρόνο χωρίς την νομοθετική βάση βρισκόμαστε στο χάος. Απαντήσω στην τελευταία ερώτηση της Προεδρού και του κυρίου Ρικέ και επίσης θα επεκταθώ στο θέμα του τομέα των αερομεταφορών για την ύπαρξη δημιουργών συμφωνιών ή την, την απουσία αυτών. Το σημερινό σύστημα ε, βασίζεται στην εξή ε, αρχή, ότι δηλαδή κάθε αεροπορική εταιρεία μπορεί ελεύθερα να πετά από ένα ευρωπαϊκό αεροδρόμιο σε άλλο. Μια αεροπορική εταιρεία ορίζεται ως ε, μια εταιρεία όπου τον έλεγχο και την ιδιοκτησία έχει στην κατοχή του κάποιος ευρωπαίος φορέας ή κάποιο ευρωπαϊκός δημόσιος φορέας κάποιου κράτους μέλους. Τώρα, no deal και plan B. Plan B. Η, πραγματικότητα μας δείχνει ότι αυτοί οι οποίοι είναι έτοιμοι για το Plan B είναι οι ιδιωτικοί φορείς, αλλά όχι οι δημόσιοι και κυρίως οι ιδιωτικοί φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, με την έννοια ότι δηλαδή οι ε, βρετανικές αεροπορικές μεταφορές, οι περισσότερες, έχουν μετατραπεί σε ευρωπαϊκές ε, εταιρείε η πλειοψηφία των μετοχών ήταν βρετανικές παλιότερα, ενώ τώρα έχουν μεταφερθεί σε μη βρετανικές εταιρείε, αλλά των 27 κρατών μελών. Άρα οι βρετανικές αεροπορικές εταιρείε, το Plan B ήταν, θα συνεχίσουμε να είμαστε ε, ευρω... ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείε. Το πρόβλημα όμως θα είναι ότι οι εταιρείε των 27 δεν θα μπορούν ελεύθερα να πετούν προς το Ηνωμένο Βασίλειο, Ελήψη συμφωνίας. Τι θα γίνει λοιπόν στην πράξη. Ή θα πρέπει να υπάρξει κάποια συμφωνία διμερής, δηλαδή η ε- Ευρώπη των 27 με το Ηνωμένο Βασίλειο και γι' αυτό βέβαια χρειάζεται χρόνος, αλλά υπάρχουν πρότυπα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συνάψει παρόμοιες ε, συμφωνίες με μη κράτη-μέλη, το Μαρόκο ας πούμε είναι το τελευταίο, η Βραζιλία είναι μια άλλη χώρα και η Άρα δηλαδή δεν ξεκινάμε από το μηδέν, διότι τέτοια πρότυπα για σύναψη συμφωνιών ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των αεροπορικών εταιριών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, της ε, θα πρέπει να σημάνει λοιπόν όπως είπαμε μια συμφωνία αλλά πρέπει να περάσει από όλη τη διαδικασία διαβούλευσης στην Ευρωπαϊκή δηλαδή θέλει χρόνο. Τώρα για τις περιφέρειες ναι, θα ήθελα να σας απαντήσω σε αυτό κυρία ε, Πρόεδρε. Όντως διαπιστώσαμε ότι η Βόρεια Γαλλία θα αντιμετωπίσει προβλήματα. Τρεις ε, ε, περιφέρειες συγκεκριμένα, Ωπ' η Νορμανδία και η Βρετάνη. Γιατί προηγουμένως είπαμε πώς ε, η ναυσιπλοεία και το κανάλι της μάχη, συγγνώμη, η σύραγγα της μάχης είναι τα πιο, οι πιο σημαντικές δίωδοι όσον αφορά το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Οπότε, ναι, εντοπίσαμε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα για τις τρεις αυτές τις περιφέρειες που βεβαίως θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε και μάλιστα στις μελέτες που κάναμε τις ε, περιπτωσιολογικές μελέτες που κάναμε ανάκρατος μελέτες για τη Γαλλία θα βρείτε αυτές τις ε, ε, πληροφορίες. Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν? Όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ε, την σύνταξη αυτής της μελέτης που σίγουρα θα βοηθήσει ώστε να δείξουμε πως οι συνέπειες ανυπαρξία συμφωνίας μπορεί να είναι καταστροφικές και μπορεί να, έχουν, να έχει αυτό αντίκτυπο σε διάφορες περιφόρειες της Ευρώπης ανάλογα με τον τομέα. Ας πούμε για τα ναυτοκινητοβιομηχανία, στις μεταφορές θα είναι πάλι τρομερές οι επιπτώσεις. Δεν το έχουμε συζητήσει τόσο αναλυτικά, αλλά και εκεί θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Ευχαριστώ για την πολύ ωραία σας παρουσίαση, πολύ ε, περιστατωμένη, όχι αισιόδοξη, αλλά μας υποχρεώνει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, ώστε να προβλέψουμε όσο γίνεται καλύτερα την κατάσταση. Μπράβο σας λοιπόν και ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μελέτη. Εγώ θα σας χειροκροτήσω και αν θέλετε και οι υπόλοιποι.